Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome to today's AFET Committee meeting. I'd like to welcome... Καλώς ορίσατε, να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνεδρίαση και να σας πω ότι περνάμε ήδη στην έγκριση της σημερινής ένταξης να σας ενημερώσω για τα εξή σημεία. Η ψηφοφορία για σήμερα το απόγευμα στο 8 σε ό,τι αφορά την ε, αυτή τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα αναβληθεί. Θα σα ανακοινώσουμε την ημερομηνία, την ψηφοφορία την επόμενη φορά και αυτό μετά από την έλλειψη, λόγω τη έλλειψη τη ε, σημαντική αυτή τη ψηφοφορία ε, και όλων των είχαν συζητηθεί 14 Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια από πλευρά σα. Η σημερινή ημερήσια διάταξη θεωρείται εγκεκριμένη. Στο 2. Δεν έχω ανακοινώσει να σα κάνω ω πρόεδρο. Στο 3. Αν δεν έχουμε σχόλια μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της συνεδρίασης 20 της 1 27η και 22 η Νοεμβρίου και 4 η Φεβρουαρίου ε, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και μετά περνάμε στο 4. Και θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Μαρία Φερνάντα Σπινόζα Γκαρσές, η οποία κάθε δίπλα μου. Είναι πρόεδρος της 73ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Εμένων Εθνών. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην ε, συνεδρίασή μας, στην Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα και με χαρά σας έχουμε μαζί μας. Η συνεργασία μεταξύ των ε, Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μακρά στην παράδοση και αυτό είναι προφανές μιας και οι δύο οργανώσεις αυτές ε, ασπάζονται και προσυπογράφουν τι αρχές και από πλευρά της Επιτροπής μας έχουμε διατρανώσει με σαφήνεια το γεγονός ότι χρειάζεται πιο στενή συνεργασία για την ε, προώθηση των προτεραιοτήτων μας, δεδομένου και το γεγονότος ότι σήμερα έχουμε δυστυχώς μεγάλες προκλήσεις για την πολυμερία. Θα προωθούμε λοιπόν την πολυμερία όπου μπορούμε και θέλουμε να συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω την υφιστάμενη συνεργασία. Και άρα, κυρία ε, Σπινόσα Γκαρσές, με χαρά θα ακούσουμε τις εργασίες σας, ε, τις ανακοινώσεις σας, τις απόψεις σας και τις προτεραιότητές σας σε ό,τι αφορά την 73η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Εθνών. Να καλωσορίσουμε και ένα τακτικό επισκέπτη της Επιτροπής μας, τον πρέσβη μας στην ε, Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι πάντα ευπρόσδεκτος ε, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Καλώς ήρθες, Ζωάο. Έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Thank you, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε της Επιτροπής αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, David, για την πρόσκληση να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας. Συχνά αναφέρομαι στη Γενική ε, Συνέλευση ως το πιο αντιπροσωπευτικό όργανο ε, το ΟΗΕ και ως το Κοινοβούλιο της Ανθρωπότητας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν να είμαι στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όχι μόνο επειδή έχουμε ζωτική σημασία σχέσεις που είναι στη δική σας αρμοδιότητα, αλλά και επειδή είστε εχμή του δόρατος της πολυμερού συνεργασίας στην πράξη για θέματα ασφάλειας, ειρήνης, απειλών ε, στο κράτος δικαίου και για το πώς συμμετέχει η Ευρώπη ε, στον κόσμο μας που είναι όλο και πιο ταραγμένος. Αγαπητοί φίλοι, είναι πολλές οι προκλήσεις, περισσεύουν και για τα δύο κοινοβούλια μας. Ε, αλλαγή, εξτρεμισμός, ε, διάδοση όπλων, ε, αλλαγή στη δυναμική των παγκοσμίων δυνάμεων και θα μπορούσα να συνεχίσω και να συνεχίζω. Με δύο λόγια είναι δυναμικές οι προκλήσεις γιατί ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και έχουμε ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο με πολλά, πολλά από τα παλιά προβλήματα να παραμένουν ενώ αναδύονται νέες προκλήσεις και προβλήματα. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκαν για να δίνουν στα κράτη καλύτερες ευκαιρίες να αντιμετωπίζουν τέτοιες απειλές και να υλοποιούν τις προσδοκίες των πολιτών τους και των ε, κρατών που τα απαρτίζουν σε συνεργασία πάντα αγαστή τη στιγμή που η πολυμερής ε, προσέγγιση αμφισβητείται, θα πρέπει να εστιάσουμε στα όσα επιτύχαμε για να απαντήσουμε στο παρόν και στο μέλλον. Παρά τις προκλήσεις λοιπόν και τα προβλήματα, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει λαμπρό φωτεινό παράδειγμα ε, του επιτεύγματος ε, κρατών όταν συνεργάζονται. Το ίδιο και για τα Ηνωμένα Έθνη. Με όλες τις αδυναμίες του ΟΗΕ έχουν, ε, έχει μετατρέψει το κόσμο σε ένα καλύτερο κόσμο. Μειώνεται η ακραία φτώχεια, ε, υιοθετούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σαλβαδόρ, ας πούμε, έχουμε από ε, στράτευση κάποιων ενόπλων και στο Νότιο Σουδάν καθαρίζουμε τις νάρκες, την αποναρκοθέτηση. Ε, πάντα η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν παραστάτης και στο πλευρό του ΟΗΕ για τη διαμεσολάβηση, την ειρήνευση, καθώς επίσης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων ε, της βίας. Έχουμε όμως και κοινά μέλη Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπων που είδαν τη ζωή τους να βελτιώνεται λόγω της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά καθώς συνεχίζεται ο πόνος και τα δεινά στη Συρία και στην Ιεμένη, ε, φαίνεται κατάφορα και ξεκάθαρα ότι απέχουμε πόρο από το κοινό μας όραμα για την ειρήνη. Κατακτήσεις που με κόπο επιτύχαμε τα περασμένα έτη τώρα αμφισβητούνται περισσότερο από ποτέ τα τελευταία 30 χρόνια. Επιθέσεις κατά των αμάχων έχουν αυξηθεί πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία. Περίπου 70 εκατομμύρια είναι εκείνοι ε, που έχουν εγκαταλείψει τις ε, αιστείες τους για να φύγουν από την πείνα, ε, από το λοιμό, από τον πόλεμο, τις βόμβες και τις διώξεις. Δεν μπορεί, όχι μια χώρα, μια περιοχή, περιφέρεια μόνη της να τα βγάλει πέρα. Είναι σαφές ότι χρειάζεται πολυμερή συνεργασία και αυτό είναι ε, επίγον. Αυτό το λέει ε, παγίως η δική μου Προεδρία και το επαναλαμβάνει. Και αυτή τη στιγμή διώκεται και υφίσταται πιέσει η πολυμερή συνεργασία. Πολλέ κυβερνήσει αναδιπλώνονται, περιχαρακώνονται, γιατί έχουν πολλά ιστορικά προβλήματα και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τα παγκόσμια. Επίση, άλλοι προσπαθούν να υπονομεύσουν την παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνε και χάνουν την εμπιστοσύνη του και την πίστη του ότι μπορούν οι οργανισμοί και οι θεσμοί να βελτιώσουν τι ζωέ του και πραγματικά χαίρομαι ε, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει προτεραιότητα για την 73η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτό το θέμα της πολυμερούς συνεργασίας. Και ως πρόεδρος κατά κάποιο τρόπο είμαι και θεματοφύλακας ε, της συλλογική προσέγγισης του συλλογικού συμφέροντος των 193 μελών των ΗΕ. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, καμιά φορά σας ζηλεύω που έχετε μόνο 28 κράτη-μέλη να βολέψετε. Γελάω. Έτσι. Κατανοώ πόσο δύσκολο είναι και με 28 κράτη και για σας Πρόεδρε, αλλά αυτή είναι η μορφιά των πολυμερών οργανισμών. Ε, δεν απειλούν την κυριαρχία των κρατών μελών. Το αντίθετο, την ενισχύουν με ενίσχυση της δυνατότητας των κρατών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν σημασία για αυτά, μοιραζόμενα το κόστος και το βάρος και ε, συνεργαζόμενα για τις βασικές παγκόσμιες προκλήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργάζονται ακριβώ προ το στόχο αυτό. Και η Γενική Συνέλευση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ηγηθούν στην προσπάθεια αυτή. Γενική Συνέλευση αντανακλά την παγκόσμια κοινή γνώμη και το βάρος της γιατί δίνει σε κάθε κράτος μέλος ε, μία έδρα, μία ψήφο και ένα μικρόφωνο. Εσείς, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι, ε, είστε οι καλύτεροι για να διαβάσετε αυτό το μήνυμα στους ε, ψηφοφόρους σας. Και φροντίζουμε και εσείς φροντίζετε συλλογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθείτε την πολυμερή συνεργασία. Δεν αρκεί όμω να λέμε ωραία λόγια για αυτή τη συνεργασία. Ο κόσμο τι θέλει. Αυτά αποτελέσματα χειροπιαστά. Εξού και το θεματολόγιο για το 2030. Είναι τόσο σημαντικό τώρα που η καιροί είναι επικίνδυνη. Καμία περιφέρεια δεν ε, είναι εμβολιασμένη και άνοση απέναντι σε ταραχές και αστάθεια. Ε, υπάρχουν υποκείμενοι λόγοι και αίτια και στα Ηνωμένα Έθνη μπορούν όλες οι κυβερνήσεις να εκφράζουν ε, τις ε, ανησυχίες τους και να πείθουν και τους πιο επιφυλακτικούς ή ε, διστακτικούς πολίτες. Έχουμε γόνιμο έδαφος τώρα για το, την άνοδο του λαϊκισμού και του εθνικισμού που επιτίθενται στην πολυμερή συνεργασία. Γι' αυτό εγώ επικεντρώνομαι ε, στην ε, αξιοπρεπή εργασία. Γιατί εκεί ε, υπάρχει πρόβλημα. Το μέλλον της εργασίας, κοινωνική προστασία, κοινωνική κινητικότητα. Αυτά είναι τα θέματα που ενώνουν τους λαούς. Για να εφαρμόσουμε απολύτως τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να δημιουργήσουμε 600 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για νέους. Ελπίζω οι χώρε σα να συμμετέχουν στη συνάντηση υψηλού επίπεδου που φιλοξενώ για την αξιοπρεπή εργασία και το μέλλον τη εργασία στι 10 του Απριλίου ε, ε, στη Νέα Υόρκη. Και πραγματικά θέλω να επενέσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσήλωσή της στους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ιδιαίτερα ό,τι αφορά τη μείωση του, χρέους, το εμπόριο και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια υπάρχει και μια ε, δημοσίευση ε, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, ακριβώς για να διαδίδονται και να φωτίζονται τα παραδείγματα καλών και βελτίστων πρακτικών. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, συνάδελφοι. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ. Το Δεκέμβριο εγκρίναμε τα σχετικά κείμενα ε, για την συντεταγμένη και ε, νόμιμη μετανάστευση. Όταν ανέλαβα, μία από τις προτεραιότητές μου ήταν να εξασφαλίσω την υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης για τα δύο αυτά σύμφωνα, και για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Ήταν μεγάλο επίτευγμα το γεγονό ότι καταφέραμε να ενώσουμε κράτη ε, για το θέμα αυτό. Μπορεί κανείς να διαφωνεί για το σύμφωνο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Υπάρχουν διστάμενε απόψει. και το κατανοώ. Όταν ήμουν στον Ισημερινό υπουργό Εξωτερικών είχα πρόσφυγε από την Κολομβία να ε, διαχειριστώ και κατανοώ πόσο σημαντικό είναι αυτό και σε εσωτερικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Αλλά η πολυμήρια συνεργασία τι σημαίνει. Να συνεχίζουμε τη συνεργασία μα και τη συζήτηση ακόμα και όταν διαφωνούμε. Για το λόγο αυτό διοργάνωσα μια συζήτηση υψηλού επίπεδου για τη διεθνή μετανάστευση και την ανάπτυξη την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και γι' αυτό το λόγο συνεργάζομαι στενά με του πρέσβει της Ισπανίας και του Μπαγκλαντές στη Νέα Υόρκη για την πρώτη αναθεώρηση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση το 2022. Αγαπητοί φίλοι, για να είμαστε πιστικοί στην πολυμερή συνεργασία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζονται διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Οι οργανισμοί μας θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικοί και να λογοδοτούν περισσότερο στους πολίτες που υπηρετούμε με ιδιαίτερη χαρά βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί προτεραιότητα ε, τη μεταρρύθμιση του συστήματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ελπίζω και εσείς ως βουλευτές να αγωνιστείτε, ε, να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζωογονηθεί η Γενική Συνέλευση και με τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλεία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η κοινωνία των πολιτών και κυρίω οι νέοι και οι γυναίκε θα συμμετέχουν ενεργά στο έργο μας να δρομολογήσουμε καλύτερα και να εξυγχρονίσουμε τις μεθόδους εργασίας. Μόνο έτσι θα έρθει πιο κοντά στον κόσμο. Χρειάζεται να διευκολύνεται για να υπάρχει η πολιτική βούληση, έτσι ώστε τα Ηνωμένα Έθνη να είναι σημαντικά για όλους. Οι νέοι υπήρξαν οι εμπνευστές των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης ανέλαβαν ε, την ε, ηγετική αυτή στάση που, που έχουν υιοθετήσει και βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώνουν στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες, σε πρωτεύουσε παντού στον κόσμο. Εγώ είμαι μόλις η τέταρτη γυναίκα στην ιστορία των 73 ετών του ΕΕ που ε, υπηρετώ ως πρόεδρο στη Γενική Συνέλευση και η πρώτη γυναίκα από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Δεν θα εκπλαγείτε λοιπόν που η ισότητα των φύλων είναι ένα θέμα για μένα ιδιαίτερα προσφυλές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντικός, κρίσιμος εταίρος των ΗΕ σε αυτό το τομέα και ε, υπολογίζω στα μέλη και προσβλέπω να μιλήσουν τα μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα ε, την Παγκοσμία ημέρα των γυναικών στη Νέα Υόρκη. Για να μην υποχωρούν τα δικαιώματα των γυναικών, ελπίζω όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης να συμμετέχουν στις 12 Μαρτίου στην διοργάνωση μας υψηλού επίπεδου που φωτίζει την θέση των γυναικών στις ηγετικέ θέσει και χαίρομαι που οι πρόεδροι της Κροατίας, Εστονίας και Λιθουανίας θα συμμετέχουν, όπως και είπατε εκπρόσωπο, η κυρία Φιντερίκα Μογκερίνη. Αγαπητοί φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κοινού στόχου για την ασφάλεια, την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την βιώσιμη ανάπτυξη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει εδώ για να προωθήσει αυτού του στόχου εντάσσοντας τα ψηφίσματα και τις αρχές του ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και εξασφαλίζοντας ε, την ταχύτερη και καλύτερη ε, εφαρμογή διεθνών συμφωνιών. Μπορείτε εσείς να ανοίξετε το δρόμο. Ας πούμε η επαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσεως είναι καταπληκτικό παράδειγμα. Αυτό που εσείς ψηφίσατε και προωθεί την παγκόσμια ε, καμπάνια για τη μείωση των πλαστικών που ξεκίνησε πέρσι. Επίσης θέλω να τονίσω ε, τη δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Θα πρέπει όλοι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να συγκρατήσουμε την κλιματική αλλαγή και την μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για να βοηθήσουμε τον Νότο, ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις μικρές νησιωτικές χώρες που χρειάζονται προσαρμογή και ε, δημιουργία δομών έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά στις νέες κλιματικές αλλαγές. Αυτό αφορά και τις επόμενες γενναίες. Και στις 28 Μαρτίου θα υποδεχτώ στη Νέα Υόρκη τη σχετική διοργάνωση. Βεβαίως έχουμε και κοινά προβλήματα και προκλήσεις. Θέλουμε οι οργανισμοί μας να είναι πιο διαφανείς και να λογοδοτούν περισσότερο. Ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέλω να φέρω τον ΟΗΕ πιο κοντά στους ανθρώπους και εσείς ως βουλευτές το ίδιο ε, επιθυμείτε και προσδοκάτε να φέρετε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες που εκπροσωπείτε. Μπορούμε να άλληλο υποστηριχθούμε ζητώντας στεναρά την πολυμερή συνεργασία. Όχι οποιαδήποτε πολυμέρεια, αλλά ε, εκείνη που θα ανταποκρίνεται, θα αποδίδει και δεν θα είναι απλώς το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων που θα έχει προστιθέμενη αξία στις παγκόσμιες ε, κρίσεις που είναι πολλές εξασφαλίζοντας ότι στην καρδιά όλων όσων κάνουμε είναι πάντα ο άνθρωπος. Με χαρά θα συζητήσω αυτά τα θέματα μαζί σας ε, σε περισσότερες λεπτομέρειες και θα είμαστε σε συνεχή επαφή για το διάλογο μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια και την εισαγωγή. Συγκρίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ε, Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών. Η διαφορά είναι ότι εμείς είμαστε απευθείας δημοκρατικά ελεγμένοι και όπως γνωρίζετε τις επόμενες εκλογές θα τις έχουμε τέλη Μαΐου που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κλίμακα δημοκρατική διαδικασία μετά τις εκλογές στην Ινδία στον κόσμο. Σε μία ενία εκλογική διαδικασία είναι πάρα πολλοί πολίτε ε, που έχουν δικαίωμα συμμετοχή. Λοιπόν, έχουμε περί τα 20-25 λεπτά χρόνο. Πρίντα, Παντζέρι, Λόχπιλα, Σούλτς, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανέναν. Αυτού έχω σημειώσει τον κατάλογο. Α ακούσουμε αυτού και μετά να ολοκληρώσουμε. Κρίστιαν Πρίντα, παρακαλώ, από το ΕΛΚΑ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, κυρία Πρόεδρο που είναι μαζί μας σήμερα. Ε, είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέρον να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με τους ε, διπλωμάτες, με τους αρμοδίους των Ηνωμένων Εθνών. Ήθελα να σας ζητήσω ή δυνατόν μία ίσως ενδελεχέστερη ανάλυση της κρίσεως τις οποίες διέρχεται η πολυμέρεια. Διότι όλο και περισσότερο αναφερόμαστε στην κρίση της πολυμέρειας και εσείς βλέπετε κάποιες αιτίε γι' αυτό. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες ε, όταν λέτε ότι η Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών είναι το, η βουλή του πλανήτη διότι οι βουλές ε, αποτελούνται από μέλη εκλεγμένα. Και επίσης μιλούμε ε, για κοινοβούλια, δηλαδή για μέρη στα οποία προασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ελευθερίες λείπουν από πολλές από τις χώρες που εκπροσωπούνται στα Ηνωμένα Έθνη. Τέλος πάντων, εσείς θεωρείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα Ηνωμένα Έθνη ε, χρησιμεύει στην χρηστή λειτουργία για παράδειγμα της υποστήριξης του καθεστώτος της Κούβας, λέει ο καθεστώς το οποίο δεν σέβεται καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε λαοτίζει πολίτες ε, λόγω των φρονημάτων τους. Επομένως, μια τόσο ευρία υποστήριξη που εκφράζει το Σώμα των Ηνωμένων Εθνών για το κουβανικό καθεστώς είναι θετικό θετικό στοιχείο για τις, ε, ε, ε, για τους φορείς και τις ε, υπηρεσίες των ΗΠΑ. Ευχαριστούμε, Κρίστιαν. Ο κύριος Παντζέρη έχει τώρα το λόγο, ε, ο οποίος θα μιλήσει Ιταλικά, λέει ο πρόεδρος. Καταλαβαίνετε εσείς Ιταλικά. Buongiorno. Καλημέρα, λέει ο μιλητής στα Ιταλικά προφανώς. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα και με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω εγώ ότι έχετε βάλει στο κέντρο της τοποθετησής σας το θέμα της ε, και της πολυπολικότητας προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες επικρίσεις που έχουν ακούσει μεταξύ άλλων από την Αμερικανική κυβέρνηση κατά των θεσμών της πολυμερίας. Εγώ νομίζω ότι η δική σας προάσπιση της προσέγγισης αυτής είναι δίκαιη και σωστή διότι η αποδυνάμωση του πολυμερού συστήματος που μέχρι σήμερα υπήρξε εγγύηση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τη συνεργασία, της ε, ανάπτυξης περαιτέρω συμφωνιών, της, του περιορισμού των συγκρούσεων, ε, είναι για μας ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Είπατε επίση, βέβαια ότι πρέπει να υποστηρίζουμε την πολυμέρεια ασκώντας επικοδομητική κριτική και επομένως προκειμένου να μην επικρατήσει η προσέγγιση και η πολιτική του πιο δυνατού που δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να οδηγεί σε συγκρούσεις πολεμικές Μήπως πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στην μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης απόφασης των Ηνωμένων Εθνών, διότι φαντάζεται κανείς πόσο δύσκολο είναι για έναν πολυμερή φορέα να λάβει αποφάσεις και τότε οδηγούμαστε σε άλλες κατευθύνσεις. Δεύτερον, η Ολομέλεια του ΟΗΕ ε, ανακοίνωσε και την δεκαετία Μαντέλα για την ειρήνη. Αυτή η δεκαετία, αυτή μάλλον την δεκαετία, καθότι ο στόχος της ειρήνης είναι θεμελιώδης, πώς θα χρησιμοποιηθεί, πώς θα αξιοποιηθεί, ώστε πραγματικά να έχουμε μια δεκαετία μεγάλης δραστηριότητας ε, υπερασπίζοντας την ειρήνη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Παντζέρη. Η κυρία Λόχπίλα για τους πρασίνους. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Εσπινόσα για την ε, εξαιρετικά ενεργητική της ηγεσία και την φιλική της ηγεσία την εκτιμούμε. Ο διάλογος υψηλού επίπεδου για το Global Compact την περασμένη εβδομάδα ήταν εξαιρετικά χρήσιμος και επιτυχής. Νομίζω ότι χρειάζεται να παρακολουθήσουμε στενά και τα δύο παγκόσμια αυτά σύμφωνα μέχρι να έχουμε κάποιες πρώτες πιο απτές ενδείξεις το 2022 για το θέμα της πολυμέρειας. Θα λέγατε ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολυμέρειας θα μπορούσαν να ενισχυθούν κάποιες συμμαχίες ή το γεφύρωμα του χάσματος βορρά-νότου, για παράδειγμα, ώστε να κινηθούμε προς τα εμπρός και ότι έτσι τελικά θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το σύστημα της πολυμερίας. Και τέλος για τα θέματα προϋπολογισμού δεν αναφερθήκατε ιδιαίτερα σε αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να επεξεργαστείτε λίγο περαιτέρω τα θέματα προϋπολογισμού του Ηνωμένων Εθνών, τα οποία νομίζω ότι θα έρθουν πολύ σύντομα φέτος ε, στο τραπέζι. Ευχαριστώ πολύ και στους όλους έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Πρόεδρο που ήλθε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ε, μιλήσατε για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το σύστημα της πολυμέρειας. Εδώ, εδώ, από τα αριστερά σας. Όπως και αρμόζει. Και εκτιμώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι είσαστε δραστήρια α, πολιτικός και σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και είσαστε πλέον ε, πρόεδρος της ε, συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα και τα τελικά βήματα για την υλοποίηση της ατζέντα του 2030 και των ε, βιώσιμων στόχων. Γιατί προφανώς όλα αυτά είναι αλληλοσυνδεόμενα. Μιλάμε για τη φτώχεια, μιλάμε για την ειρήνη, την ενίσχυση των περιβαλλοντικών πτυχών, το καθαρό νερό, το οποίο αποτελεί βασική αναγκαιότητα για δισεκατομμύρια ανθρώπους παντού. Άρα, η Γενική Συνέλευση, ο ΙΕ, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να πετύχουν τους στόχους αυτούς. Τι πιθανότητες υπάρχουν και ύστερα μία άλλη ερώτηση σε ό,τι αφορά και τις ε, πολύ δύσκολες εποχές που περνάμε στην ε, Ευρώπη, σε ό,τι αφορά την ε, ακύρωση της συνθήκης για τους πυράβλους Μεσογλυνικούς. Βρισκόμαστε σε έναν διαρκες διαρκές πινκ-πονκ μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτών. Και θα αναφέρουμε και τον ελέφαντα στην αίθουσα. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να επανέλθουμε σε ένα καθεστώς ε, πυρηνικής, ε, πυρηνικού αφοπλισμού προκειμένου και η νέα γενιά να έχει την αισιοδοξία για το μέλλον. Και είναι πολύ ενισχυτικό το γεγονό το ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Washington Post δημοσίευσε ένα άρθρο για, για κρυφή επιστημονική έρευνα για τον ιό της γρήπης. ένα είδος δηλαδή βιολογικού όπλου. Και αυτό επανέρχεται ως θέμα στην Ευρώπη, Ευρώπη γιατί η ΕΠΑ μαζί με τις κατοχώρες ε, αναπτύσσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει ετοιμότητα στο σύστημα του ΟΗΕ για να υπάρξει αντίσταση σε αυτές τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα νέα αυτά όπλα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, συναδελφοί, δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Και γι' αυτό λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Κοιτάξτε, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις πολύ επίκαιρες αυτές και πολύ ε, σωστέ ερωτήσει. Το πιο βασικό νομίζω έχει να κάνει με το πώ μπορούμε να ενισχύσουμε την πολυμέρια. και γιατί το λέμε ξανά και ξανά ότι η πολυμέρια είναι υπό επίθεση. Απειλείται. Γιατί λοιπόν. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα παράδοξο. Ζούμε σε έναν κόσμο όλο και πιο συνδεδεμένο και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι όσο το επιτοπλίστων διεθνικές προκλήσεις που δεν γνωρίζουν σύνορα το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, η αλλαγή του κλίματος, το θέμα του πυρηνικού εξοπλισμού, η πυρηνική απειλή, η τρομοκρατία. Όλες αυτές οι προκλήσεις δεν έχουν να κάνουν με μία και μόνο χώρα. Απειλούν όλη την ανθρωπότητα και είναι αν θέλετε και προκλήσεις που απειλούν την ίδια μας την επιβίωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο ισχυρή, πιο οργανωμένη πολυμερία, πιο πολλή συνεργασία, πιο πολλές συλλογικές δράσεις και θα πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει πραγματικά η κοινή ευθύνη. Όλα αυτά λοιπόν μας εξωθούν σε ένα σύστημα πολυμέρειας και μια τάξη βάσει κανόνων και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει από κοινού να ταχθούμε υπέρ της πολυμερίας. Και όπως σας είπα, δεν χρειαζόμαστε όποια πολυμέρεια μα έλθει στο κεφάλι, αλλά χρειαζόμαστε μια πολυμέρεια η οποία θα εξυπηρετεί το στόχο για τον οποίο έχει καταρτιστεί. Γιατί δεν είναι η στιγμή να χάσουμε την εμπιστοσύνη μα στι πολυμερεί αυτέ ε, οργανώσει. Γιατί όμω υπάρχει αυτή η απώλεια εμπιστοσύνη, Γιατί καταρχά χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία από κοινού, συλλογικά. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει να υπάρξουν πιο πολλά συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι το πιο ισχυρό εργαλείο που καταδεικνύει ότι πραγματικά είμαστε σε θέση να πετύχουμε τους στόχους μας είναι η, στόχη, η βιώσιμη στόχη της Αυτοί νομίζω καταδεικνύουν κατεξοχήν το τι μπορεί να πετύχει το πολυμερές σύστημα Σήμερα λοιπόν αντιμετωπίζουμε την πρόκληση αυτή και όπω είπε ο κ. έχουμε την ευκαιρία να αγγίξουμε πραγματικά τη ζωή του κάθε πολίτη και αυτό το έχουν κατανοήσει τα Ηνωμένα Έθνη και γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε στην παρούσα φάση να ξεκινήσουμε μία εκβάθρον διαδικασία μεταρρύθμιση. Κάνουμε μεταρρύθμιση λοιπόν αναθεώρηση και επανεξέταση του συστήματός μας σε τρεις βασικούς πυλώνες. Αλλάζουμε όλο το οικοδόμημα τις οργανωσές μας και το θέμα της ανάπτυξης και το θέμα της ασφάλειας και της ειρήνης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί πιο πολύ η αρχή της επικουρικότητας, να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και προφανώς είμαστε σε μια διαδικασία μεταρρύθμισης της όλης, ε, του όλου συστήματος διαχείρισης. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Θα δούμε λοιπόν τι θα πετύχουμε και τι θα καταφέρουμε ως οργάνωση μέσω της αναθεώρησης αυτής. Ένα άλλο ζήτημα. Ο ρόλος μας ως οργάνωση πρόληψης των συγκρούσεων. Εδώ νομίζω ότι έχουμε πετύχει πολλά εργαζόμαστε υπό την αρχή της διατήρησης της ειρήνης. Η αρχή λοιπόν αυτή βασίζεται στην προληπτική αυτή διάσταση. Έγινε ένα ερώτημα για τη δεκαετία της ειρήνης. Εμείς επιμένουμε και επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση της ειρήνης. Η ιδέα λοιπόν αυτή συνδέεται προφανώς με την εφαρμογή της ατζέντα το 2030 και τους βιώσιμους στόχους. Επίσης, ετέθησε ένα ερώτημα για τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και πώς μπορούμε να πετύχουμε μια συμμαχία καινούρια. Ελπίζω να μην επαναλαμβάνομαι υπερβολικά, αλλά νομίζω ότι όταν μιλάμε για την κρίζωση της φτώχειας, των ανισοτήτων, όταν μιλάμε για την ατζέντα για την αλλαγή του κλίματος. Όλα αυτά αποτελούν κοινού παρανομαστές και για τον ε, Βορρά και για τον Νότο. Δεν βλέπω γιατί η αλλαγή του κλίματος αφορά μόνο τον Νότο. Είναι στην ατζέντα όλων. Όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των διαστατικών αιτιών της ε, φτώχειας ε, και της, του αποκλεισμού Μιλάμε για κοινή ατζέντα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να γίνει διάκριση τεχνητή μεταξύ βορρά και νότου. Το θέμα είναι η ανθρωπότητα σε όλον τον πλανήτη να είναι σε καλύτερη θέση. Και αυτό προασπίζεται ο ΙΕ ως οργάνωση. Και προφανώς ε, ως ε, μια ανθρωπογενής οργάνωση έχουμε πολλές προκλήσεις πάντα να αντιμετωπίσουμε. Οι προκλήσεις όμως αυτές θεωρώ ότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική βούληση των κρατών μελών. Καταλαβαίνω πολύ καλά ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κοινοβουλίου που συναποτελείται από α, ε, ερετούς βουλευτές και μιας οργάνωσης ε, που απαρτίζεται από μέλη κυβερνήσεων και έχουν διοριστεί από κυβερνήσεις οι οποίες πάλι έχουν εκλεχθεί. Είμαστε λοιπόν, έχουμε προσώπους από 93 χώρες και θα πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Έχουμε τις κοινέ αρχές και τους κοινούς στόχους προς εφαρμογή και είναι πραγματικά πολύ φιλοδοξή η ατζέντα μας. <coughs> Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για να ωφεληθούν τελικά τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν εκδιωχθεί από τη χώρα προέλευσής τους. Το θέμα της πυρηνικής απειλής, ε, του GPCOA και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις ε, σε ό,τι αφορά και την πολυμέρεια είναι να υπάρξει ένα διεθνές σύστημα βάσει κανόνων. Θα πρέπει αυτό να το προωθήσουμε. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας, τα νομοθετήματα που έχουμε προσυπογράψει και με μεγάλη μου ικανοποίηση είτε και την τοποθέτηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Και, αν δεν κάνω λάθος, αυτές ήταν οι ερωτήσεις που μου θέσατε. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άλλος συνάδελφος έχει καμιά ερώτηση, καμιά αναπάντητη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι στις Βρυξέλλες θα έχετε και άλλες ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Πότε γυρνάτε στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα πάω στο Ελσίνκι. Okay. So, good luck, good success. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και στο καλό να πάτε. Λοιπόν, μπορούμε τώρα συνάδελφοι να περάσουμε περίπου στην ώρα μας το επόμενο θέμα. Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή παρακολούθησης των εκλογών στη Μολδαβία στις 24 Φεβρουαρίου. Θα θυμάστε ότι ε, στο τελευταίο ψήφισμα για τη Μολδαβία που εγκρίθηκε πέρσι τον Νοέμβρη, επαναλάβαμε τη θέση μας και παραθέτω οποιαδήποτε απόφαση για μελλοντική μακροοικονομική εκταμείευση ε, θα λάβει χώρα μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές και υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει σύμφωνα με διεθνώς αναγορισμένες προδιαγραφές και θα αξιολογηθεί από τους αρμόδιους φορείς και το πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης ε, θα παραμείνει σε αναμονή μέχρι να υπάρξει η μετάβαση ε, και η αλλαγή στη χώρα. Και τέλος της ε, παρέμφεσης. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αξιολόγηση από ανεξάρτητους παρατηρητές για τις μελλοντικές σχέσεις με τη Μολδαβία. Πενταμελής επιτροπή ορίστηκε που εκπροσωπούν τέσσερις πολιτικές ομάδες ε, με πρόεδρο την κυρία Ρεμπέκα Χάρμς και μακροπρόθεσμα εγγράφεται στις αποστολέ ΟΑΣΕ και ΟΔΙΡ και του Συμβουλίου τη Ευρώπη σύμφωνα με τι ε, διεθνεί αυστηρέ προδιαγραφέ και μεθοδολογία του ΟΑΣΕ ΟΔΙΡ. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Ρεπέκα Χάρμς, επικεφαλής αντιπροσωπεία, για να μα ε, πει πώ αξιολογεί τι εκλογέ. Και θυμίζω, συνάδελφε, ότι στις 4 και 4 αναμένουμε τον Πρωθυπουργό τη Αρμενία. Δηλαδή ακριβώ 30 λεπτά και λιγότερο έχουμε για το θέμα αυτό. Παρακαλώ Ρεμπόκα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, και τα μέλη του προσωπικού της αντιπροσωπείας μας. Ήταν πάρα πολύ καλή επιστολή, πολύ καλό το κλίμα εργασίας. Ε, μια χώρα που είναι αρκετά περίπλοκη έτσι, πολιτικά και οι συνθήκες που επικρατούν εκεί στη Μολδαβία. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους των πολιτικών ομάδων, το προσωπικό που μας βοήθησε να λύσουμε το πρόβλημα μια δεύτερη ε, ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε εγγραφεί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τελικά μετά από εντατικές ανταλλαγές και συνεννοήσεις μεταξύ μας στη Μολδαβία, ε, συνεννοήσεις με τις υπηρεσίες των Βρυξελών και με τη βοήθεια του πρέσβη μας στο Κίσενάου, η δεύτερη εναλλακτική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν κατέφτασε στη χώρα και καλά έκανε. Γιατί αυτό βοήθησε να πετύχει η δική μας αποστολή ε, ε, μετά από αυτή την αγαστή συνεργασία ε, Κίσενάου και Βρυξελών. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την Κριστίνα. Τι κάναμε λοιπόν εκεί που πήγαμε. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε διάφορους ενδιαφερομένους που εκπροσωπούν διάφορα πολιτικά κόμματα, μέσα ενημέρωσης και ΜΚΟ. Επίσης, βασιστήκαμε στα βρήματα κάποιων άλλων παρατηρητών έτσι πιο μακροπρόθεσμο. Δεν θέλω να επεκταθώ. Υπήρχαν κάποια προβληματικά στοιχεία ε, ε, για άνηση ε, πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης από κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίσης, ακούσαμε παράπονα και διαμαρτυρίες για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και ισχυρές καταγγελίες για την κατάχρηση εξουσίας. Ποιο είναι το πρόβλημα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αντιπροσωπεία μας δηλαδή, αλλά και εκείνη του ΟΝΤΙΡ, του ΟΑΣΕ, περιέγραψαν τις εκλογές της 24ης Φεβρουαρίου ως ανταγωνιστικές. Είχαμε την αίσθηση ότι έγιναν με τρόπο επαγγελματικό τα διαδικαστικά, δηλαδή τα εκλογικά τμήματα είχαν καλή διαχείριση, κυρίως γυναίκες ήταν οι πρόεδροι. 40% ε, είναι ε, η ποσόστοση που προβλέπεται για τις γυναίκες υποψήφιες, οι οποίες ήταν 40% αλλά όχι σε εκλόγιμες θέσεις, σε πολύ χαμηλή θέση στο ψηφοδέλτιο. Οι εκλογές αυτές επίσης ε, θεωρήθηκαν ως τεστ, δοκιμή για να περιφερωθεί η εκταμείευση της μακροοικονομικής βοήθειας, αλλά και για το μέλλον των σχέσεών μας και της συνεργασίας μας και την εύρυθμη λειτουργία της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλά αρνητικά τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή μας. Και επίσης το αναφέρουμε ρητά και στη δήλωσή μας και το είπαμε και εκεί την επομένη των εκλογών στο Κεσινάου συμμετοχή κάτω από το μισό των εγγεγραμμένων σε εκλογικούς καταλόγους, πολύ χαμηλότερο από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το 2014, αλλά και στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών το 2016, τα μεγαλύτερη αποχή λοιπόν. Αυτό μάλλον οφείλεται στη μείωση της εμπιστοσύνης και της πίστης ε, του πληθυσμού ε, στους δημόσιους φορείς και στις αρχές λόγω των αρνητικών εξελίξεων που είχαμε μετά το 2014 και τις εκλογές του 2014. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στην τεράστια τραπεζική απάτη το 2014 η οποία ακόμα είναι υποδιερεύνηση. Αργεί η δικαιοσύνη και οι διαδικασίες στα δικαστήρια ε, για εκείνους που έχουν ανοιχνευτεί ε, ε, και ο Ιλάν Σόρ, α πούμε, που ήταν στην υπόθεση της απάτης, κατέβηκε στι εκλογές με το κόμμα που είχε το όνομά του, το κόμμα του Σόρ, που βγήκε τέταρτο στις εκλογές, στι βουλευτικές. Ακύρωση επίσης ε, των εκλογών του 2018 για το Δήμο του Κεσινάου. Επίσης είναι ένα από τα αρνητικά στοιχεία και αρνητική εμπειρία για τους ψηφοφόρους. Επίσης υπάρχει μεγάλη διαπλοκή ολιγαρχών με πολιτικούς και έχει αλλάξει η σύνθεση του, ε, του Κοινοβουλίου της χώρας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Ήταν και μεικτό το σύστημα για τις βουλευτικές εκλογές Εγκρίθηκε το, στα μέσα του 2018 ο νέος εκλογικός ε, νόμος χωρίς διαβούλευση δημόσια ε, και χωρίς αποκλεισμούς. Και αυτό το έχει ε, επικρίνει και η Επιτροπή της Βενετίας και ο ΑΣΕ και ο ΝΤΙΡ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμά του του 2018. Μπορεί να το θυμάστε. «50 βουλευτές έχουν, ένα σώμα έχει βουλή με αναλογική με εθνικά ψηφοδέλτια. Και έχουν νέες μονοεδρικές 51 ε, περιφέρειες. Έχει γίνει κατάχρηση εξουσίας, κατάχρηση δημοσίου χρήματος με πίεση των δημοσίων υπαλλήλων να ψηφίσουν. Ε, και με έλεγχο των μέσων ενημέρωσης που δεν παρουσιάζουν όλες τις απόψεις τους ψηφοφόρους. Ε, ήταν κάπως συγκεχημένη η κατάσταση γενικώ και κατά την άποψή μας ε, εσκεμένα. Ε, ήταν τέσσερα διαφορετικά τα ψηφοδέλτια που έπρεπε να βάλει κανείς στην ίδια κάλπη για την εθνική επικράτεια, για τις μονοεδρικές και για δύο μη δεσμευτικά δημοψηφίσματα που έγιναν όλα ταυτόχρονα με τις βουλευτικές εκλογές. Το είδαμε αυτό σε διάφορα εκλογικά τμήματα. Ο κόσμος είχε μπερδευτεί, δεν ήξερε τι ψήφισε. Επίσης, είδαμε και κάποιες ε, αναντιστοιχίες ή μάλλον κάποια, παράβαση του απορρίτου των, ε, της εκλογικής διαδικασίας και Επίσης υπήρξε μεγάλη διακριτική μεταχείριση βάρος των Μολδαβών που δεν ζουν στη Μολδαβία που δεν μπορούσαν να ψηφίσουν μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ενώ εκείνοι που ζουν στη Μολδαβία μπορούσαν. Όσοι ζουν στη διασπορά, στο εξωτερικό και έχει λήξει το διαβατήριό τους, δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν, σε αντίθεση με τα όσα έγιναν το 2014 και το 2016, όπου τότε ψήφιζαν και με λιγμένα διαβατήρια. Και μόνο στις 14 Ιανουαρίου η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξέρετε αν έχετε λιγμένο διαβατήριο δεν πρόκειται να το δεχτούμε για να ψηφίσετε. Και αυτό δυσκόλευε. Τους πολίτες δεν προλάβανε να βγάλουν καινούριο διαβατήριο για να ψηφίσουν. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση ε, το ε, που δέχτηκαν πολλοί πολίτες από την υπερνηστερία που δεν τους άφηναν να ψηφίσουν ή άλλους τους ε, ε, ε, είχαν καταγγείλει ότι χρηματίστηκαν και είχαν διοργανωθεί μαζικές μεταφορές τους για να ψηφίσουν. Μεγάλη γενοδορία λοιπόν επέδειξε η κυβέρνηση για πολίτες που ζουν ε, σε περιοχέ χώρες που δεν ελέγχονται από την κρατική και κεντρική κυβέρνηση. Τελειώνω, τελειώνω. Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν τα τρία μεγάλα κόμματα, οι σοσιαλιστές, οι δημοκράτες και το μπλοκ ΑΚΟΥΜ, ε, πήραν 27 και 34 έδρε από τις 101 αυτό δείχνει τώρα ότι είναι δύσκολο να σχηματιστεί η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, και γιατί έχουν κάνει δηλώσει οι ηγέτε των τριών μεγάλων κομμάτων κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εξαρτία ότι μεταξύ του δεν συνεργάζονται. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, προβλέπονται ε, νέε εκλογέ σε 4 με πέντε μήνε. Τα υπόλοιπα προβλήματα τα γνωρίζετε πολύ καλά και τα έχουμε συζητήσει και μάλιστα επανειλημμένα στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Χάρμς για την ε, εκτεταμένη αυτή η ανάλυση σχετικά με την αποστολή της 24ης Φεβρουαρίου. Έχουμε περί τα 15 λεπτά τώρα για ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πρέντα, Κριστέα, Πώς, Οστρεβίτσιους, Τσέλα, Μούντι. και Γκόμες. Επτά ομιλητές, ε, δύο λεπτά έκαστος. Παρακαλώ. Κύριε Πρέντα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Ρεμπέκα Χάρμς. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η διαδικασία δεν συνιστούν κάποια βελτίωση δημοκρατική, όπως ίσως ελπίζαμε, αλλά είναι μια επιβεβαίωση των προσπαθειών του Κοινοβουλίου μετά την επίκριση της Επιτροπής Βενετίας για το νέο αυτό εκλογικό νόμο, εκλογικό σύστημα, το οποίο δεν επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση των πολιτών, αλλά έχουμε κάποιους ε, ημετέρους, ε, κάποιους που πρόσκυνται στο Κρεμλίνο, κάποιους ε, όχι κτλ. Δεύτερον, η ψήφος στην Τρασινιστρία, στην Υπερνιστρία, είναι υπό τον ολιγάρχη Πλαχόντνικ ε, φοβούμε πως αυτοί οι ίδιοι οι ψηφοφόροι θα χρησιμοποιηθούν γιατί έχουν και ε, διαβατήρια ρουμανικά και ίσως να τα χρησιμοποιήσουν για εκλογές κράτους μέλους, δηλαδή του δικού μου. Ε, εν η ψήφο στην υπερνιστρία ενέχει ένα σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Τρίτον, νομίζω ότι όχι μόνο πρέπει να αναστείλουμε την ενίσχυση, την δημοσιονομική, αλλά πρέπει να καταδείξουμε όλους εκείνους τους άρχες ε, που είναι υπεύθυνοι για τη διαφθορά, υποστηρίζουν το καθεστώς 100%, ελέγχουν το καθεστώς απολύτως, ε, και το καθοδηγούν σε συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες είναι στην άμεση γειτονία μας. Ε, πρέπει να περάσουμε λοιπόν σε μια στάση πιο στεναρή και δεν πρέπει να υποκύψουμε στους εκβιασμούς ε, που δεχόμαστε από το καθεστώς. Ευχαριστούμε, Κρίστιαν, ευχαριστούμε για τα δύο λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γεωπολιτικός μιλώντας, η η δημοκρατία της Μολδαβίας υπήρξε πάντοτε σημαντική στην περίπτωση των εκλογών. Για παράδειγμα το 2014. Είχαμε μια δυτικόστροφη ε, κυβέρνηση. Αν δει κανείς πώς το πράγμα οργανώνεται αυτή τη στιγμή, διαρθρώνεται αυτή τη στιγμή, είχαμε την επιβεβαίωση των επικρίσεων του μεικτού συστήματος που είχαμε νωρίτερα. Τα πράγματα πρέπει ακόμα να βελτιωθούν, αλλά εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγει τις εκλογές. Είχαμε μια συμφωνία σύνδεσης με συγκεκριμένα σημεία και κεφάλαια. Τα, τα υφιστάμενα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο έχει διαρρεθεί, κάποια κόμματα είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Υπάρχουν άμεσες διασυνδέσεις ε, με το L και το SND ε, μάλιστα, αλλά πρέπει να δούμε κατά πόσον θα τοποθετήσουν το δικό του συμφέρον πρώτα. Εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά τις δικές μας επιλογές, διότι ίσως να υπάρξει και μια υποβάθμιση της ε, πολιτικής ανατολικής γειτονίας και διαρωτώ με τι θα γίνει με τη Μολδαβία, όπου έχουμε αυτό το διαρρεμένο κοινοβούλιο και ίσως να δούμε το ίδιο και στην Ουκρανία, λέει ο μιλητής. Έχουμε Σελίνσκι, Τιμοσέγκο, Ποροσέγκο, την, ε, το τριμερές αυτό σχήμα. Ε, αλλά θα είμαστε ρεαλιστές ε, με το Κισίνεφ ή θα έχουμε μία στάση άσε να δούμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καθόλου κατάλληλο κάτι τέτοιο. Πρέπει να είμαστε προδραστικοί και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη που έχουμε και ιδιαίτερα οι πολιτικές ομάδες που ενέχονται. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αουστρεβίτσιους, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλει σαφή μηνύματα για την ε, δημοσιονομική υποστήριξη στα πλαίσια της Συμφωνίας ε, Σύνδεσης. Εκτιμώ την ε, έκθεση της Ρεμπέκα και την εμπειρογνωμοσύνη της στο ζήτημα και την εμπειρία που είχε. Ακούμε κάποιες θετικές και κάποιες αρνητικές αναλύσεις. Εγώ ως εισηγητής της ΑΦΕΤ και ω μέλος πολιτικής ομάδας που δεν έχει καμία σχέση με τα ε, πολιτικά κόμματα που μόλι εξελέγησαν στο ε, Κοινοβούλιο τη Μολδαβία, θα έλεγα ότι η εικόνα δεν είναι ούτε απολύτω λευκή, ούτε απολύτω μελανή. Η, καταρχάς η εκλογική διαδικασία δεν έχει απολύτω τερματιστεί, ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κάποιε διαδικασίε προσφυγής οι οποίε ακόμα είναι εν εξελίξη και ίσω να χρειαστούν περί τι 7 εβδομάδε για να έχουμε τις τελικές εκθέσεις των αρμοδίων. Ε, επομένως, ε, Πρόεδρε, θα έλεγα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή δεν θα πρέπει πρόημα να αξιολογήσουν την διαδικασία των εκλογών και τις σχέσεις με τη χώρα αυτή. Και το λέω αυτό διότι είμαι βέβαιος ότι το 2017 λάβαμε μια πολύ σωστή απόφαση και διαθεσμικά μάλιστα ε, και θα έμενα στο πλαίσιο και στην κατεύθυνση της συμφωνίας εκείνης για να δω την τελική έκθεση, τα τελικά πορίσματα. Θα πρέπει να δούμε πώς η μολδαβική κυβέρνηση θα χειριστεί όλες αυτές τις ε, καταγγελίες και τις προσφυγές και ίσως να είναι αποφασιστικός παραγών. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους αυτούς που συμμετείχαν στην ε, αποστολή παρακολούθησης. Τσέλα, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το πόσο διαφορετικέ είναι οι εντυπώσει ε, για τι εκλογέ αυτέ ε, είναι σαφέ από το, το γεγονό ότι η κυρία Χάραμ μα παρουσίασε ένα μεγάλο κατάλογο για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Σε, ενώ, για παράδειγμα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ε, δήλωσε ότι όλα πήγαν εξαιρετικά, δίκαια και κανένα πρόβλημα πόσο διαφορετικά λοιπόν μπορούμε να εκτιμούμε διαφορετικέ καταστάσει. Αυτό που διαπιστώνουμε ωστόσο είναι ότι μειώθηκε έτσι περαιτέρω η προσέλευση στι κάλπε στη Μολδαβία κάτω από 50% πλέον. Και το μοναδικό θετικό θεωρώ είναι ότι ο συνασπισμό ε, τη αντιπολίτευση ε, εξακολουθεί να έχει 27 έδρε στο Κοινοβούλιο. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πληρωμή, για την αναστολή μάλλον των πληρωμών σε ό,τι αφορά την ε, δικαστική μεταρρύθμιση ήταν σωστή. Μιας και δεν υπάρχει καμία πρόεδρος εκεί και ανακοινώθηκε ότι πριν την ε, σύσταση στη σώμα του Κοινοβουλίου θα μεταβεί στην Μόσχα για να συνομιλήσει με τον ε, πρόεδρο Πούτιν και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία Κανένα κυβερνητικό σχηματισμό με τη συμμετοχή του κόμματος ΣΟΑ και ότι οι διαφορέ είναι τόσο μεγάλε που δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο νέων εκλογών. Εγώ ήμουν σε μια περιοχή όπου είχαμε πολλούς από την υπερνηστερία και είχαμε ειδικά εκλογικά κέντρα για τους ανθρώπους αυτούς, για τους πολίτες αυτούς από τις 11 λοιπόν το πρωί άρχισαν να καταφτάνουν ε, τα πούλμαν. Όταν τους μιλούσαμε στη γλώσσα τους, ε, ε, μας απαντούσαν αμέσως, στα ρωσικά σιωπούσαν αμέσως και δεν έδινε, δεν έδινε καμία απάντηση. Στο Κισινάου δεν υπήρχαν ε, τέτοια εκλογικά κέντρα και εκεί ήμουν στο τέλος της εκλογικής διαδικασίας. Ε, έκανα μια παραγγελία σε ένα μαγαζί, ζήτησα να πάρω κάτι και η κυρία εκεί στο μαγαζί μου είπε ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ τόσους πολλούς ρωσόφωνους <laughs> με... να έρχονται και να πληρώνουν με μεγάλα νομίσματα. Με 100 λέει. Έχουμε λοιπόν την συμφωνία σύνδεση με την Μολδαβία αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της κατάστασης εκεί και πραγματικά την υποστήριξή μας θα πρέπει να την δώσουμε στις πραγματικά, στην πραγματική αντιπολίτευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μύρος Λαφμπός, ευχαριστούμε κύριε Τσέλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ συμμετείχα στην αντιπροσωπή αυτή. Οι εκλογέ ήταν ελεύθερε και δίκαιε. παρά το γεγονό ότι στην προεκλογική εκστρατεία είχαμε προβλήματα και ακόμα νιώθαμε τον αντίκτυπο των εκλογών στο Κισνάου πέρσι. Ήταν ελεύθερε οι εκλογέ και παρά το γεγονό ότι νίκησε το κόμμα το ρωσικό των Ρώσων, τα αποτελέσματα ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι περι... περιμέναμε. Δεν έχουμε ε, λαϊκιστές, δεν έχουμε κομμουνιστές, άρα παρά την μαζική προπαγάνδα που επικρατούσε, η κατάσταση στη Μολδαβία φαίνεται ότι είναι καλύτερη από όταν στο παρελθόν. Χαίρομαι, ε, μάλλον λυπάμαι που το κόμμα υπέρ της Ευρώπης σημείωσε μάλλον οριακά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά και τη συμμετοχή σε ένα συνασπισμό. Γιατί θεωρώ ότι διαφορετικά η κατάσταση ήταν διαφορετική. Ακούσαμε μεγάλη κριτική σε ό,τι αφορά το σύστημα των εκλογών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή της Βενετίας, όλα αυτά. Πιστεύω ότι αποτέλεσαν ε, με έναν τρόπο να μπουν στην ε, πολιτική σκηνή της Μολδαβίας νέες δυνάμεις. από τις συγκεκριμένες ε, περιοχές. Η εξαρτία λοιπόν δεν είχε να κάνει μόνο με γεωπολιτικά ζητήματα μεγάλης κλίμακας, αλλά και με τοπικά ζητήματα. Να πω δύο λόγια, γιατί εγώ ήμουν στην, ε, στο Νότο, στην αυτόνομη περιοχή του Κάφκασου και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο κύμα επενδύσεων από την Τουρκία και εδώ θα πρέπει να εστιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μόντι και μετά η κυρία Γκόμες. Mm. Σας ευχαριστώ πολύ και είναι ενδιαφέρον που ακούμε τις εντυπώσεις των προηγούμενων μελητών που ήταν παρόντες ε, και έτσι αυτό μας δίνει και μία εντύπωση για το πόσο απλό θα είναι να δημιουργηθεί συνασπισμός. Ήταν τόσο ανταγωνιστικές άλλωστε οι προεκλογικέ του εκστρατείε. και αν δεν καταφέρουν να σχηματίσουν συνασπισμό, τι διαφορά θα κάνουν νέε ερωτήσει ή νέε εκλογέ. Δεύτερη ερώτηση. Πώ μπορούμε εμεί να δραματίσουμε επικοδομητικό ρόλο στην πολιτική της Μολδαβίας παρά να περιοριστούμε στην κριτική. Θέλω λοιπόν να είμαστε πιο επικοδομητικοί στη στάση μας και να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τη Μολδαβία στην επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κλέρ, και τέλος να ακούσουμε και την Ανά Γκόμες. Και περιμένει ήδη έξω ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας. Ναι, συγγνώμη, λέει η κυρία Γκόμες. Εγώ δεν ήμουν στην αποστολή, αλλά με ανησύχησε η έκθεση της κυρίας Ρεμπέκα Χάρμς. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τόσοι πολλοί πολίτες δεν κατέβηκαν στις εκλογές. Ακόμα και ο ΑΣΕ αναγνωρίζει το πρόβλημα αυτό. Και νομίζω ότι σε κάποιε περιπτώσει είχαμε και ακύρωση εκλογών σε περιπτώσει που δεν υπήρχε επαρκή προσέλευση. Συμφωνώ το ερώτημα τη Κλέρ Μούντι προ την ε, Ρεμπέκα. Πώ μπορούμε να αντιδραματίσουμε επικοδομητικό ρόλο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρο τι αρχέ μα. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τον κόσμο στη Μολδαβία και αν θέλουμε να βοηθήσουμε και του εαυτού μα στην τελική ανάλυση. Right, uh, ευχαριστώ. Ρεμπέκα, κοίτα να δεις. πιέζει το πρωτόκολλο. Αν είναι ένα λεπτό, ένα λεπτό και ούτε λεπτό παραπάνω. Πιστεύω λοιπόν, εξ όσων κατάλαβα, πολλοί πολίτες στη Μολδαβία κατάλαβαν και εκείνοι τι κάναμε όταν βάλαμε όρους για την εκταμείευση της μακροοικονομικής βοήθειας, τους οποίους δεν θα πρέπει να αλλάξουμε. Δεύτερον, Ό,τι και να κάνουμε, και ό,τι και αν κάνουμε, που θα πρέπει να το αποφασίσουμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να είμαστε συνένοχοι στη μεγάλη διαφθορά. Ευχαριστώ πολύ, ε, Ρεμπέκα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν έχουμε χρόνο για μεγαλύτερη συζήτηση και ζητώ και συγγνώμη από τους εκπροσώπους της ΑΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι τη Ρεμπέκα Χάρμς και όλους τους συναδέλφους που πήγαν εκεί στην αποστολή παρατήρησης των εκλογών και είμαι βέβαιος ότι η χώρα αυτή θα εξακολουθεί να μας απασχολεί εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων χωρίς καμιά αμφιβολία. Ωραία. Ολοκληρώνεται το σημείο 5. Μια στιγμή πάω να υποδεχτώ τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like... Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, να συνεχίσουμε με το σημείο 6 τη Μεσσίας διατάξεω. Είναι χαρά και τιμή μα να υποδεχόμαστε τον κύριο Νικόλ Πασινιάν, Πρωθυπουργό τη Ερμενίας, για ανταλλαγή απόψεων. Πρωθυπουργέ, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα που όπω λέτε και στην γλώσσα σα μπάρει γκαλός, αν το λέω καλά, Καλώ ήλθατε. Νομίζω ένα χειροκρότημα το αξίζει ο Πρωθυπουργό. And I have now honor... Και έχω την τιμή να υποδεχθώ και άλλους προσκεκλημένους από την Αρμενία. Και έχω το, την τεράστια πρόκληση της προφοράς των ονομάτων τους. Δίπλα στον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μενατσακιάν, αναπληρωτής πρωθυπουργός Μέρ Γκριγκόριαν ε, καλώς ήλθατε ο Υπουργός Παιδείας Αράρικ Χαρουτουμιάν αν το λέμε καλά καλώς ήλθατε όλοι οι προσκεκλημένοι είναι τιμή όπως έλεγα Πρωθυπουργέ που σας δεχόμαστε εδώ σήμερα μετά το πολύ θερμό, τη θερμή φιλοξενία πέρυσι, όπου είχαμε πάει στις 18 Ιουνίου, μετά την επίσκεψη ε, αυτή είχαμε τις ε, πιο σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις με ειρηνικές διαδηλώσεις που κατέληξαν ε, στην πρωθυπουργοποίησή σας σε ένα πρόγραμμα εντολή κατά της διαφθοράς κυρίως. Μετά σημειώσατε και σημαντική νίκη στις εκλογές τις κοινοβουλευτικές και η κυρία Χάουτολα, η συνάδελφος, παρατήρησε από την αποστολή ότι οι εκλογές αυτές ήταν καλά διοργανωμένες, με πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις παρατυπίας και υψηλό επίπεδο εγγυήσεων. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν που βρίσκεστε εδώ. Έχετε το λόγο βεβαίως Πρωθυπουργέ και ελπίζω να έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους συναδέλφου. Να σας θυμίσω όμως ότι στα, σε 55 περίπου λεπτά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την συνάντηση αυτή γιατί έχουμε και άλλα θέματα στη διάταξη. Παρακαλώ Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε Μακάλιστερ. Επτά μέλη, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τιμή και χαρά μου που απευθύνομαι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι μετά την ειρηνική μας εξέγερση είναι η πρώτη ευκαιρία για τον Πρωθυπουργό να απευθύνεται στην ΑΦΕΤ. Θα ήθελα λοιπόν να εστιαστώ ιδιαίτερα στις θεμελιακές αλλαγές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μου. Θα ήθελα να μιλήσω και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα όπως και για τους στόχους και σχέδιά μας για το μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Αρμενία διέρχεται σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών άνευ προηγουμένου στην κλίμακά τους και τα οποία μεταμορφώνουν απολύτως το πολιτικό και οικονομικό μας πεδίο, σκηνικό. Την περασμένη άνοιξη είχαμε μια ειρηνική επανάσταση όπου οι πολίτες με συνθήματα την αγάπη και την αλληλεγγύη ύψωσαν το ανάστημά τους για να οικοδομήσουμε μια κοινωνία που να είναι σύμφωνη προς τα ιδεώδη των πολιτών. Ε, προτίμησαν τον πλουραλισμό και την δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ισότητα και κατέκριναν την διαφθορά και ένα πελατειακό κομματικό σύστημα που είχαμε προηγουμένως και τάχθηκαν κατά της ελίτ των, της οικονομικής και της πολιτικής που είχαμε, της, του ολιγαρχικού συστήματος οικονομίας, κατά εκείνων που εκμεταλλεύονταν τους θεσμούς οδηγώντας την χώρα σε τέλμα. Η Επανάσταση η Βελούδινη αποκατέστησε την δημοκρατία και είχαμε τις εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου που ενίσχυσαν τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα της επανάστασης αυτής. Ε, σημειώσαμε ευρύτατη νίκη και οι πολίτες ε, εξέφρασαν σε πάνω από 70% των ψήφων την υποστήριξή τους. Για πρώτη φορά σε 25 χρόνια οι εκλογές της Ερμενίας δεν αμφισβητήθηκαν από κανένα πολιτικό κόμμα. Είναι εξίσου σημαντικό να πούμε ότι η πρόσφατη εκλογική διαδικασία είχε την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση από τους παρατηρητές Ευρωπαϊκής Ένωσης που την θεώρησαν, τις θεώρησαν ελεύθερες και δίκαιες. Η νίκη της δημοκρατίας είναι πλέον ε, αδιαφυσβήτητη και μη μεταστρέψιμη στη χώρα μας επί των εξής αξώνων. Η δημοκρατία και η ισότητα είναι πλέον εγγεγραμμένη στο γενετικό κώδικα των πολιτών και της κοινωνίας. Η Αρμενία ήταν από τις πρώτες χώρες όπου είχαμε ένα κοινωνικό κίνημα, λαϊκό κίνημα, ήδη από τη δεκαετία του 80, η αποκατάσταση δημοκρατίας το 1991, αδιαφυσβήτητα προσπαθούσε να οικοδομήσει την κοινωνία επί τη βάση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Η διαστρέβλωση της δημοκρατίας που είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια έλαβε χώρα ως αποτέλεσμα αποκλήσεων από, τον, από την αρχική κατεύθυνση που είχαμε επιλέξει και προήλθε από μια λανθασμένη και παραπλανητική ερμηνεία των αξιών και ιδεωδών μας η δημοκρατική μεταμόρφωση της κοινωνίας μας βασίζεται σε, μια ευρύτατη, σε ένα ευρύτατο κοινωνικό αίτημα από, όλα, από όλες τις κοινωνικές ομάδες και των 6 εκατομμυρίων βεβαίως της αρμενικής διασποράς παγκοσμίω και ε, ανέκυψε ως φιλοδοξία και αίτημα του λαού των πολιτών δεν είχε καμία σχέση με εξωτερικά κέντρα ή δυνάμεις και δεν προκάλεσε καμία τεκτονική αλλαγή στις εξωτερικές μας σχέσεις ούτε στην στρατηγική την εξωτερική μας. Μένουμε δεσμευμένοι στις εξωτερικές μας σχέσεις και τους εταίρους μας. Η δημοκρατία βεβαίως δεν είναι απλώς μία από τις επιλογές που είχαμε μπροστά μας. Είναι θέμα επιβίωσης και ασφάλειας για εμάς. Θεωρούμε ότι στην παράδοση και τον πολιτισμό μας η δημοκρατία είναι το μόνο σύστημα που παρέχει ισχυρότερες οικονομικές και κοινωνικές δομές που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας χώρας. Δεν μπορούσαμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να έχουμε την πολυτέλεια των ημιτελών προηγουμένων θεσμών που είχαμε στη χώρα που παρεμπόδιζαν την οικονομική μεγέθυνση και την πρόοδό μας. Η προώθηση των οικονομικών και πολιτικών μας θεσμών ήταν απολύτως απαραίτητη. Δεν υπήρξε καμία, δεν είχαμε καμία εναλλακτική λύση, εκτός από τη δημοκρατία, για να εισέλθουμε και εμείς τον 21ο αιώνα τελικά. Και πρέπει να ενισχύσει το δημοκρατικό σύστημα και να αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις που έχουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα την ένδια που ακόμα υπάρχει στη χώρα. Οι πολίτες που ζουν υπό το όριο της ένδυας είναι περί το 1 τρίτο του πληθυσμού. Και είναι η βασική πηγή της διαφθοράς και της ε, απάτης ε, της εκλογικής που είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχει ένας προφανής συσχετισμός μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της δημοκρατίας. Η αποδόμηση της μέσης τάξης ήταν η αιτία της υποχώρησης της δημοκρατικής που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως μια ισχυρή και βιώσιμη μέση τάξη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της επιβίωσης και ενίσχυσης δημοκρατίας. Ο επόμενος λοιπόν στόχος της κυβέρνησής μας και ακρογωνίος λόθος, του προγραμματός μας είναι αυτός. Και με αυτό κατά νου υιοθετήσαμε και ήδη εφαρμόζουμε μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα θεματολόγιο μεταρρύθμισης και μεταξύ των ε, υφισταμένων προτεραιοτήτων της ε, αρμενικής κυβέρνηση έχουμε τον πόλεμο κατά τη διαφθορά, την εκρίζωση των μονοπωλίων, την αντιμετώπιση της φτώχεια, την ε, εγκατάσταση και υποστήριξη ενός ανεξαρτήτου συστήματος δικαιοσύνη και ένα σύστημα ισότιμο και δίκαιο για όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς θα προχωρήσουμε σε, ένα, σε μια δέσμη μέτρο για την μεταρρύθμιση, την φορολογική και των τελωνίων. Θα προχωρήσουμε στην μεταρρύθμιση του ζητήματος παιδείας, διότι οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε έναν συνεχώς μεταλλασσόμενο κόσμο, πλανήτη, που οθείται από τη γνώση. Είμαι υπερήφανος που σας ανακοινώνω ότι πολλές αλλαγές απτές και εμφανείς ήδη έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας. Για παράδειγμα, εκριζώσαμε ήδη την συστηματική διαφθορά που αντιμετωπίζαμε. Η δύναμη των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων μετριάστηκε σημαντικά. Σήμερα κανείς στην Αρμενία δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει, να ασκήσει πολιτική επιρροή για να επιτύχει οικονομικούς στόχους. Εφαρμόζοντας την εξωτερική μας πολιτική, αγαπητοί συνάδελφοι, αντιμετωπίζουμε ακόμα εμπόδια και ένα πράγμα είναι απολύτως σαφές. Η υλοποίηση της ε, ευρύτατης συμφωνία σύνδεσης εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, είναι θεμελιώδης για την πρόοδό μας. Και εδώ πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας αποκλειστικά μέσω της υλοποίηση μεταρρυθμιστικών μέσων, μέτρων. Η υλοποίηση των μέτρων αυτών θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές σε πολλά πεδία της κοινωνίας μας, σε πολλούς τομείς και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση της Αρμενίας είναι απολύτως αποφασισμένη να εκτελέσει και να υλοποιήσει όλα τα μέτρα της, της συμφωνίας αυτής προκειμένου να έχουμε μια καρποφόρο συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κοινά επίπεδα ενδιαφέροντος, συμφέροντος. Η επικύρωση λοιπόν της ΕΠΑ από τα κράτη-μέλη θα ήθελα να θυμίσω ότι είναι κρίσιμης σημασίας για την απόλυτη θέση σε ισχύ της και για να ενισχύσει τις διμερείς μας σχέσεις. Στο σημείο αυτό, άνω του ενός τρίτου των κρατών μελών έχουν ήδη επικυρώσει τη συμφωνία και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Επ' αυτού πραγματικά υπολογίζουμε, βασιζόμαστε στην ε, υποστήριξη και την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο του θεματολογίου συνεργασίας μας θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην απελευθέρωση των θεωρήσεων και το σχετικό διάλογο. Το άνοιγμα αυτής διαδικασίας θα βοηθήσει τις επαφές μεταξύ των πολιτών και στην συνεργασία μας συνολικά. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας να προωθήσουμε το στόχο αυτό, καθότι η Αρμενία συστηματικά υλοποιεί όλες τις προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Η οικονομική και τεχνική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμη σημασίας για εμάς. Χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για να πραγματοποιήσουμε αποφασιστικά βήματα της μεταρρυθμιστικής μας ατζέντα. Το σύστημα της άμεσης ε, σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα προς τα εμπρός. Και όσο ταχύτερη η αρρωγή, τόσο ταχύτερη θα είναι και η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, γεωπολιτικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου, είναι μέρος των προκλήσεων και εμποδίων που αντιμετωπίζουμε, υποσκάπτουν διαρκώς το δυναμικό μας των μεταρρυθμίσεων, καταρχάς η ανεπίλητη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, με τάσεις που, με αντίκτυπο που ζούμε και στη χώρα μας. Αυτό επηρεάζει την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας και της όλης περιοχής. Δεύτερον, αυτή, αυτός ο αγώνας εξοπλισμών στον οποίο έχουν προχωρήσει οι αντίπαλοι μας είναι μια δυσκολία για τον Νότιο Κάφκασο. Η Αρμενία υποχρεούται να δαπανά σημαντικό μέρος των ε, πενιχρών της μέσων στους εξοπλισμούς που εξακολουθούν να είναι τροχοπέδι αλλά αποτρέπουν νέα ανάφλεξη των συγκρούσεων. Τα κλειστά σύνορα επίσης και το εμπάργκο που μας έχουν επιβάλει από, την, από νωρίς δεκαετία του 1990 ε, περιορίζει σημαντικά δραστικά την ε, οικονομία μας. Επίσης το σύστημα κυρώσεων ε, του Ιράν μας αστερεί τον, από τον έναν εκ των δύο διαδρόμων ε, συνεργασίας και εμπορίας που έχουμε με τον κόσμο. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, όπως καθότι αναφέρθηκα στην σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, θα ήθελα να αναφερθώ και στην πολύ ισορροπημένη και επικοδομητική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τις ειρηνευτικές ε, προσπάθειες του OSCE Minsk Group στέλνοντας το σαφές μήνυμα ότι η χρήση βίας, η χρήση των όπλων είναι απαράδεκτη. Η επίλυση της διαφοράς εξαρτάται απολύτως από την κατανόηση της ε, ανάγκης των κατοίκων του Ναγκόρνο Καραμπάχ ε, να έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Εδώ και άνω των δύο δεκαετιών ζουν σε μια de facto ανεξαρτησία οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν ε, νεαροί άνθρωποι εκεί που δεν μπορούν να φανταστούν τίποτε άλλο από την απόλυτη ανεξαρτησία. Αν θέλουμε μια ειρηνευτική τελική λύση θα πρέπει να επιτραπεί στους ε, πολίτες του Ναγκόρνου Καραμπάχ να διαμορφώσουν μόνοι τους το μέλλον τους. Δεν εκπροσωπώ βεβαίως τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Έχω μόνο την εντολή των πολιτών της Αρμενίας και όχι του αρμενικού πληθυσμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ που έχει το δικό του σύνταγμα και έχει τη δική του κυβερνητική δομή. Είναι απολύτως προφανές για μένα ότι η ειρήνευση μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον ο λαός του Ναγκόρνο Καραμπάχ εκπροσωπείται στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών. Γιατί μόνο αν ακουστεί η φωνή των κατοίκων του Ναγκόρνο Καραμπάχ θα μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. αξιότιμα μέλη είναι απεποίθησή μας απόλυτη ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών είναι μια από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την επίλυση οποιασδήποτε σύγκρουσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαλόγου και αμοιβαία κατανόησης. Εμείς βλέπουμε τον Νότιο Κάφκασο ως περιοχή όπου ανεξαρτήτως κρατών ζουν και μπορούν να ζήσουν αλληλέγγυα και σε συνεργασία διάφοροι λαοί και διάφορες χώρες. Τα κλειστά σύνορα είναι μια οικονομική ανοησία. Δεν έχουν κανένα νόημα. Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνδέσεις. Έχουμε όλο και πιο πολυεπίπεδο συσχετισμό χρειαζόμαστε μια νέα μορφή διαλόγου που να στηρίζεται στην οικονομική συνεργασία και την οικονομική ανάπτυξη. Ο διάλογος και η αλληλεγγύη και ανοχή θα πρέπει να υπερισχύουν απέναντι οποιασδήποτε άλλης διαφοράς μπορεί να υπάρχει στην περιοχή του σου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Prime Minister, thank you ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά σχόλια και νομίζω ότι πραγματικά ήταν ε, πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σα. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι και μεγάλο αριθμό των συναδέλφων που συμμετέχουν στη σημερινή μα συνεδρίαση και τη ζητούν το λόγο καταδεικνύουν και το έντονο ενδιαφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα για τη χώρα σα. Να σα υπενθυμίσω ότι συνενέσαμε στι 4 Ιουλίου για την ε, συνεκτική συμφωνία με τη συνθήκη με την Αρμενία στην Ολομέλεια, 173 ε, ψήφοι και 50 ήταν οι ψήφοι κατά και 43 οι αποχές για το θέμα των θεωρήσεων. Είπαμε στο ψήφισμα εκείνο ότι προσβλέπουμε στην απελευθέρωση, στην έναξη του διαλόγου μάλλον για την απελευθέρωση από το καθεστώς των θεωρήσεων. Φυσικά στα κράτη-μέλη επαφίεται τώρα να ξεκινήσουν το σχετικό διάλογο και προφανώ και πρέπει να υπάρξει ομοφωνία, αλλά εμεί τουλάχιστον είμαστε σαφεί στην τοποθέτησή μα, συνάδελφοι. 12 άτομα, 12 άτομα, επαναλαμβάνω, ζητούν το λόγο. Αν όλοι τηρήσετε το όριο των δύο λεπτών, θα έχουμε 25 ε, λεπτά ερωτήσει ε, και μετά θα δώσουμε 15 λεπτά στον Πρωθυπουργό του λόγο για να απαντήσει. Μάλιστα. Συμφωνείτε όλοι. Να ξεκινήσουμε με τον επικεφαλή ε, τη αντιπροσωπεία για την περιοχή αυτή, τον κύριο Σαγιάτ Καρύμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, ε, με Υπουργέ Εξωτερικών, ε, είναι μεγάλη ικανοποίηση από πλευρά τη αντιπροσωπεία μου και εξ ονόματο των συναδέλφων μου να σα καλωσορίσω εδώ σήμερα. Είναι σαφέ, όταν είχαμε συναντηθεί για πρώτη φορά, κανεί δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει αυτό το μονοπάτι, αυτή την οδό που ακολούθησε η Αρμενία και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το καλωσορίζουμε όλο ιδιαίτερο και κυρίω πάνω από όλα αυτά, πάνω θεωρώ ότι δίνει το μήνυμα της ευκαιρίας, της ευκαιρίας η οποία υποστηρίζεται απόλυτα από τη βούληση του λαού σας. Αυτό καταδεικνύεται και καταδείχθη πρόσφατα από τα εκλογικά αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, των οποίων επικεφαλής είναι η κυρία Χάουτουλα, για την συμμετοχή τους στην διαδικασία διεξαγωγή των εκλογών, το οποίο μας επιτρέπει με απόλυτη βεβαιότητα να σας απευθύνουμε τα συγχαρητήριά, τα συγχαρητήριά μας, κύριε Πρωθυπουργέ. Για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και τις σχέσεις τις οποίες διατηρούμε στην παρούσα φάση. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρία σχόλια, εν συντομία, μετά από τα εισαγωγικά μου αυτά σχόλια. Η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστια. Το τόνισε αυτό. Περιλαμβάνει για την Αρμενία μεγάλες ευκαιρίες, περιλαμβάνει και τις περιφερειακές ευκαιρίες όμως που ανοίγονται τις σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Να είστε βέβαιος κύριε Πρωθυπουργέ, όπως είπε και ο κύριος ε, πρόεδρος ο κύριος ε, Μακάλιστερ ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς το Κοινοβούλιο της Αρμενίας σε ό,τι αφορά την πρόθεση της ΕΠΑ μέσω της ε, συνεργασίας με την Αρμενία και πιστεύουμε ότι τώρα και οι υπόλοιποι θα πρέπει και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν αυτό που τους αναλογεί για να μπορέσουμε να επικυρώσουμε τη διαδικασία αυτή και να εμβαθύνουμε τις ε, σχέσεις μας όπως το επιθυμούμε εσωτερικά. Α, συγγνώμη, ξεπέρασα το χρονικό όριο, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Να κάνετε τρία σχόλια για την περιφερειακή κατάσταση τώρα. Έχετε δίκιο, κύριε Πρωθυπουργέ. Τα σύνορα παραμένουν μεν κλειστά. Οι οικονομικές ευκαιρίες ε, και η ασφάλεια της ε, Αρμενίας πολύ απλά δεν έχουν όμως την υποστήριξη που θα ήθελε ο λαός της Αρμενίας προκειμένου να υπάρξει πρόοδος και σε άλλους τομείς. Επ' αυτού θεωρώ ότι θα διαπιστώσετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει και των προηγούμενων ψηφισμάτων του θα μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει υποστηρίξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σάκη λέει ο Πρόεδρος. Να περάσουμε τώρα στους ομιλητέ από τις πολιτικές ομάδες και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τόκιο από το ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο του ομιλητή. Κάνει διακοπές. Δεν ακούγεται ο μιλητής, μάλλον πρέπει να αλλάξει μικρόφωνο. Δυστυχώ ο μιλητή δεν ακούγεται. Μιλάει σε ένα μικρόφωνο που δεν λειτουργεί. Κύριε Τόκιο, λέει ο προεδρό. νομίζω ότι το μικρόφωνο σας δεν λειτουργεί καθόλου. Τόση ώρα μιλάτε και δεν ακούγεστε. Δεν υπάρχει διερμηνία σε καμία γλώσσα γιατί δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Δεν σας ακούνε οι διερμηνείς. Μήπως να αλλάξετε θέση, να αλλάξετε μικρόφωνο. Ανάβει το φως. Ναι, το ξέρω ότι ανάβει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Μπορεί κάποιος να αποκαλεί τη χώρα του δημοκρατία και να μην είναι. Ξέρετε, δεν είσαι ότι δηλώσει πάντα. So, we are now enlightened. Please continue. Τώρα φωτιστήκαμε. Ε, παρακαλώ. Καλώς ορίζω τις θετικές εξελίξεις μετά ε, τις βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2018 και διάβασα την έκθεση των παρατηρητών εκλογών όπως παρουσίασε την έκθεση αυτή η επικεφαλής συνάδελφος κυρία Χάιντι Χάουταλα. Η χώρα μου λοιπόν στα πλαίσια αυτά, η Ρουμανία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αρμενίας και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας προς την κατεύθυνση αυτή. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες, ε, τις μεταρρυθμιστικές της χώρας, ιδιαίτερα γιατί είναι σημαντικές για τη μελλοντική συνεργασία. Και επειδή υπάρχουν θετικές εξελίξεις, πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα τώρα να θεωρήσουμε ότι μπορεί να αρχίσει ο διάλογος ή να υποστηρίξουμε την έναρξη διαλόγου για απελευθέρωση ε, θεωρήσεων διαβατήριων που έχουν λάβει ήδη οι γείτονέ σα Μολδαβία και Γεωργία. Για να γίνει όμως αυτό και να το υποστηρίξουμε υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος κριτηρίων που πρέπει ακόμα να πληρωθούν. Άρα αυτό σημαίνει ότι εσείς κύριε Πρωθυπουργέ θα πρέπει να συνεχίσετε και να ελοποιήσετε τις δεσμεύσεις που αναλάβατε ως κυβέρνηση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ε, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στις προσπάθειες εκδημοκρατισμού της χώρας σας. Ο Θεός να σας έχει καλά. Ευχαριστώ σοσιαλιστές και δημοκράτες, η Κλέρ Μούντι. Ε, welcome, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας εφηρεώνετε το χρόνο σας σήμερα το απόγευμα. Ήμουν και εγώ τμήμα, μέλος της αντιπροσωπείας ε, στο Νότιο Κάφκασο και ήμουν και μέλος της ε, Επιτροπής για την Παρακολούθηση των Εκλογών. Είναι λοιπόν χαρά μου που έχω την ευκαιρία για να σας επεκτείνω το λόγο. Τρία στοιχεία ήθελα να θίξω. Όπως επισημάνετε και εσείς ο ίδιος, έχετε μακρύ κατάλογο με όλα όσα πρέπει να γίνουν. Οι τομείς και οι προτεραιότητες οι οποίες ε, αναφέρατε για μια καλύτερη οικονομία για τον λαό της Αρμενίας, προφανώς αυτό είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων σας και το θέμα της μέσης τάξης κτλ. Θα πάρουν χρόνο όμως όλες αυτές οι ενέργειες, έτσι για να έχετε, πρέπει να διαχειριστείτε και τις προσδοκίες σας, να αναγνωρίσετε την υπομονή και την επιμονή που θα χρειαστεί η υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων αυτών. Τι σχέδια λοιπόν έχετε σε ό,τι αφορά την παρουσίαση και την διαχείριση των προσδοκιών. Κατά δεύτερον, το θέμα της είπα και το θέμα της ε, επικοινωνίας, της προώθησης ε, του θέματος αυτού ως ενός θέματος το οποίο θα είναι υπέρ του λαού της Αρμενίας. Όχι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ποια είναι η στρατηγική επικοινωνία σας προς τον λαό της Αρμενίας για το θέμα αυτό. Και τέλος, ο ρόλος των γυναικών. Η αντιπροσωπεία σας είναι μάλλον ανδροκρατούμενη και ξέρω φυσικά ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες εξαιρετικές στην Αρμενία και θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε για να αναδεχθούν πιο πολλές γυναίκες σε υψηλές ηγετικές θέσεις και στην Αρμενία. Και πάλι σας ευχαριστώ που ήλθατε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορείτε να χαλαρώσετε για 20 λεπτάκια, γιατί όλοι οι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο και νομίζω καλύτερα να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις. Απολαύστε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξαιρετικό. Από του φιλελευθέρου, ο κύριος Αουστραβίτσιος. Σας παρακαλώ, μην υπερβαίνετε τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και χαίρομαι για την επικοδομητική σας ε, προσέγγιση προς τους φιλελευθέρους, ιδιαίτερα όταν μας τριμώχνετε για το χρόνο. Ε, καλώς ορίσατε. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, Συνήθω. χαιρόμαστε πολύ να ε, συνομιλούμε με τους εταίρους μας παγκοσμίω και ιδιαίτερα από τον Νότιο Κάφκασο. Ε, τονίσατε την ειρηνική αλλαγή που επήλθε στην Αρμενία, που είναι πραγματικά εξαιρετική εξέλιξη ως πολιτική διαδικασία και γίγνεστε στη χώρα. Δεν ισχύει αυτό για όλες τις χώρες της περιοχής σας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα και πολύ γερό. Αλλά υπάρχει ένα αίσθημα δικαιοσύνης που θα πρέπει να εδρεωθεί στο λαό. Γιατί αυτές οι αλλαγές γέννησαν και μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες τώρα πρέπει να υλοποιηθούν παρακολουθήσαμε ε, σκάνδαλα διαφθοράς, αποκαλύψεις, ε, ηγέτες στο παρελθόν ε, έκλεψαν κρατική περιουσία σε επίπεδα άνευ προηγουμένου. Τι γίνεται στη δικαιοσύνη έχουν ε, προσαχθεί εκείνοι ε, που ενέχονται σε αυτά τα σκάνδαλα διαφθοράς. Υπάρχουν αυτά αποτελέσματα. Και δεύτερη ερώτηση αφορά τη γεωπολιτική κατάσταση. Πολύ σωστά είπατε ότι η Αρμενία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και προς τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Πώς θα περιγράφατε τις σημερινές σας σχέσεις με τη Ρωσία που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις εξελίξεις στην Αρμενία και θα είχατε την καλοσύνη να σχολιάσετε λίγο και τις υβριδικές απειλές ιδιαίτερα τα θέματα προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί εναντίον της χώρας σας και των πολιτικών αλλαγών. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας τύχη. Ευχαριστώ Πέτρας, ε, τους Πρασίνους ή Ρεμπέκα Χάμς, παρακαλώ. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, είχα και εγώ τη χαρά να επισκεφθώ τη χώρα σας αμέσως μετά τη Βελούδινη Επανάσταση και μετά είχα και μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση να έρθω για τις εκλογές. Και όλοι οι συνάδελφοι της αντιπροσωπείας έχουμε την αίσθηση ότι ο κόσμος περίμενε με μεγάλο ενθουσιασμό και πολλές ελπίδες στις εκλογές αυτές. Και δεν μπορούμε παρά να σας συγχαρούμε για τα όσα μέχρι τώρα έχετε επιτύχει. Ταυτόχρονα όμως παρακολουθούμε και παρατηρούμε ότι αυτός ο ενθουσιασμός, οι ελπίδες και οι προσδοκίες ε, βαρύνουν τώρα τους δικούς σας ώμους και τους ώμους κυβέρνηση, και θα ήθελα να προσπαθήσω να καταλάβω καλύτερα ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνετε πέρα από τη συμφωνία και την κύρωση της συμφωνίας ΣΕΠΑ. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα και πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την ε, καλύτερη ανάπτυξη στην Αρμενία. Και πώς θα βγάζετε πέρα με την αύξηση των τιμών φυσικού αερίου από την Gazprom αμέσως μετά την εκλογική σας νίκη. Ανέβασαν τις τιμές φυσικού αερίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάλλη από την ομάδα EFDF. Στα αγγλικά, ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κύριε Πρωθυπουργέ. Θα σας διαβάσω το κείμενο του συναδέλφου Καστάλντο που έχει άλλες ανελημμένες υποχρεώσεις και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Είναι στα Ιταλικά, οπότε σας παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Thank you. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε μια φάση πολύ σημαντική για τις σχέσεις μεταξύ Αρμενίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έδειξε και η επίσκεψη του Επιτρόπου Χάν, του πρέσβης Βιτάρσκι, αλλά και όπως ενέκρινε η Ολομέλεια πέρυσι, για την ενισχυμένη αυτή συμφωνία ΣΕΠΑ και χωρίς να αναφερθώ στις τελευταίες ε, κοινοβουλευτικές εκλογές με υψηλό δίκτυ διαφάνειας και ευθυγράμμισης με τα διεθνή πρότυπα. Όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία που είναι απλώς η αρχή μιας πορείας που θα πρέπει να περπατήσουν μαζί η Αρμενία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλος χώρα, Επιστρέφοντας στην ΣΕΠΑ, ήθελα να σας ε, ρωτήσω πώς ε, προβλέπετε να προχωρήσετε στην υλοποίησή σας. Έχω... Ε, έχουμε θετικά, θετικές ενδείξεις και σημάδια και από τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρθηκε στην δυνητική αύξηση των πόρων ενίσχυσης. Δεύτερον, ήθελα να αναφερθώ στην περίπτωση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Από την ομάδα Μίνσκ είχαμε μάθει ότι είχατε δεχθεί να συναντηθείτε. Τι περιμένετε από τη συνάντηση, από το διάλογο αυτό και με βάση τις ε, θετικές ενδείξεις από την ομάδα επαφής. Περιμένετε να έχουμε σημαντικά νέα. Θα Σα εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε πολλά να κάνετε στη χώρα σας. Είναι φιλόδοξο το πρόγραμμά σας. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια από το ΕΛΚ ο συνάδελφος Τέτινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Βάλτε σας παρακαλώ τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω τσεχικά. Καλώς ορίσατε, Πρωθυπουργέ. Αναφερθήκατε σε διάφορες εξελίξεις στη χώρα σας και πραγματικά Εκτιμώ πολύ το πολιτικό πολιτισμό των συμπολιτών σας ε, που προχώρησαν σε όλες αυτές τις αλλαγές με τόσο πολιτισμένο τρόπο. Και αυτή η επανάσταση αποκαλείται βελούδινη επανάσταση, παρχέτνα για ρεβολούτσια στα ρωσικά. Και εγώ είμαι Τσέχος ο ίδιος και χάρηκα πάρα πολύ που δανειστήκατε ε, αυτή την έκφραση από τη δική μας βελούδινη επανάσταση. Αναφερθήκατε και στη σύγκρουση για το ορεινό Καραμπάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ. ήθελα να σας πω ότι οι Αρμένοι της Επιτροπής Αρτσάχ ήταν εκείνοι που οδήγησαν ε, στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Από το 1988 ήρθαν αυτοί οι Αρμένοι στην Τσεχοσλοβακία και κατέθεσαν λουλούδια εκεί που είχε αυτοπυρποληθεί ο εθνικός μας ήρωας Γιάν Πάλαχ διαμαρτυρόμενος κατά της ε, ρωσικής εισβολής. Ήταν η πρώτη σοβιετική η Αρμένοι εκείνη που εκφράστηκαν κατά της κατοχής. Και έρχομαι στην ερώτησή μου για τη σύγκρουση στον Αγκόνο Καραμπάχ. Για ποιο λόγο η Αρμενία δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Σας ευχαριστώ για την απάντηση που θα μου δώσετε. Ευχαριστώ. Έξι ακόμα συναδέλφους έχουμε στον κατάλογο, ο οποίος και κλείνει. Η Αναγκόμες σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ορίσατε. Και θέλω να καλωσορίσω και την επανάσταση όπου πρωταγωνιστήσατε. Είμαι από την Πορτογαλία και έχουμε ειδική σχέση με την χώρα σας. Ε, γιατί έχουμε και ένα εξέχοντα Αρμένη στη χώρα μας που έκανε πολύ μεγάλη διαφορά και διακρίθηκε. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Αν θέλετε να ανακτήσετε ε, τα κλοπημαία και τα χρήματα αυτά από τη διαφθορά που έχουν μάλλον επενδυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπάρχει η Unicry που είναι ένας θεσμός που λειτουργεί εδώ στις Βρυξέλλες που μπορεί να σας βοηθήσει γιατί ακριβώς αυτή είναι η δουλειά του. Η ανάκτηση των ε, κλαπέντων ε, στοιχείων ενεργητικού από τους διεφθαρμένους ηγέτες. Από το 2003 και μετά αυτή τη δουλειά κάνουν για πολλές χώρες και με την Αραβική Άνοιξη από το 2013 και μετά. Θα μπορούσαν και για σας να το κάνουν. Υποτίθεται ότι εσείς έχετε επίσης ε, τα πιο επικίνδυνα πυρηνικά εργοστάσια στην Αρμενία και προσπάθησε συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εμπλακεί ε, στον ασφαλή παροπλισμό και αντικατάστασή τους. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε κανένα τέτοιο πρόγραμμα για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας ακριβώς για να ξεφύγετε από αυτό τον εκβιασμό που σας κάνει τώρα η Gazprom και γενικότερα στρατηγικά για, το καλό του λαού σας και ολόκληρης της περιοχής. ECR, κυρία Φωτίγκα. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Εμείς παρακολουθήσαμε, παρατηρούμε τις εξελίξεις στη χώρα σας και την κατάσταση με μεγάλη προσοχή και όσο και ενδιαφέρον μεγάλο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο ανησυχεί η Αρμενία όπως ανησυχούμε και εμείς για τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία. Δεν περιμένω μακροσκελή ομιλία, αλλά θέλω να μου πείτε αν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά. Some comments concerning... Uh, και ποιες είναι οι σχέσεις με την Τουρκία. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Η πράσινη, η κυρία Λόχμπίλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλώς ορίσατε, Πρωθυπουργέ. Στην ομιλία σας είπατε ότι η εξωτερική σας πολιτική δεν θα αλλάξει, δεν θα υπάρξουν αλλαγές και θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής. Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα ε, ε, είναι πολύ ε, απαραίτητο να ε, ενισχύσουμε το κράτος δικαίου, μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Και ε, υπό τη δική σας διακυβέρνηση, ε, καλό θα ήταν να ενισχυθεί και το διεθνές δίκαιο και η διεθνής δικαιοσύνη. Σκέφτεσαι να κυρώσετε το καθεστώς της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, ε, γιατί αυτό που περιλαμβάνεται και στη Συμφωνία Εταιρική Σχέση. Ευχαριστώ. Ο Χέρμουτ Σόλτ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω θερμά τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. προηγουμένω, ε, μιλήσατε εκτενώς για την συνεργασία και για τις δημοκρατικές εξελίξεις στη χώρα σας, για τα κοινωνικά ζητήματα, για το ε, πόσο ο λαός ε, συμμετέχει και τι γίνεται με τη φτώχεια. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα ε, για τα οικονομικά βήματα που προτίθεστε τώρα να κάνετε τα επόμενα χρόνια ή και τους επόμενους μήνες για να ξεπεραστεί αυτή η φτώχεια. Γιατί η φτώχεια μπορεί να καλλιεργήσει τη διαφθορά, είναι αποτελέσει γόνιμο έδαφος. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αρμενία αλλά και η γεωργική παραγωγή θα πληγούν από αυτή. Ευχαριστώ, Χέλμοντ Σόλτ. Ο Μιχέλ Γκάλερ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, ευχαριστώ Πρόεδρε μάλλον, ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, τον καλωσορίζω και εγώ. Αναγνωρίζουμε ότι έχετε τεράστιες προκλήσεις μπροστά σας. Η συμφωνία που μόλις ε, συνάψαμε ε, σημειώνει προσεκτικά το γεγονός ότι ε, βρίσκεστε σε αυτό σε αυτήν την Ευρασιατική Τελωνακή Ένωση. Η ερώτησή μου είναι ότι αυτή η ένωση σημαίνει ότι όλα τα αγαθά που εξάγεται προς τη Ρωσία είναι ανεφδασμών. Αυτό είναι τουλάχιστον για σας μια ελεύθερη αγορά. Αφενός. Αφετέρου, στα πλαίσια της συμφωνίας εστιαζόμαστε επίσης ή μάλλον κυρίως στα θέματα κράτους δικαίου στα οποία πρέπει να επικεντρώνεται οποιαδήποτε χώρα που βρίσκεται σε μεταβατική φάση. Ήσασταν αισιόδοξο. Ε, εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες ότι δεν υπάρχει πια καμία συστημική διαφθορά στην Αρμενία. Μακάρι να είναι έτσι. Ε, είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα φιλοδοξούσαν να αναλάβουν το κερδοφόρο αυτό πεδίο εκ νέου. Ε, είμαι σίγουρο ότι υπάρχει, υπάρχουν πειρασμοί, για να το πω έτσι και ε, καθότι είχαμε μια εμπειρία ε, στην βοήθεια, στην ενίσχυση χωρών που περνούσαν τέτοιες μεταρρυθμιστικές ε, μεταβατικές φάσεις σε τι θέλετε να επικεντρωθείτε στην μεταρρύθμιση δικαιοσύνη, των δημοσίων προ... συμβάσεων, των τελωνιακών αρχών, της Γενικής εισαγγελία, δηλαδή όλες αυτές οι δομές που είναι η παρακαταθήκη της ε, παλαιότερης κατάστασης διακυβέρνησης. Ε, σε τι από αυτά θα βλέπατε μια, ένα σημείο προτεραιότητος και στο πλαίσιο της Νέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, λέει ο Πρόεδρος. Έχω και την Heidi Hout, αλλά νομίζω. Μισό λεπτό. Charles Τάλεκ. Έτοιμα που μόλις τώρα το κάνετε δεν το κάνατε από την αρχή το έτοιμά σας να σημειωθεί. Κοιτάξτε, επειδή ε, πολύ λίγες ε, μέρες μας έχουν μείνει μέχρι τις 29 Μαρτίου, κατανοούμε τους Βρετανούς ε, συναδέλφους. Η κυρία Χάουταλα τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, ηγήθηκα δύο αποστολών παρατήρησης, ε, τον Απρίλιο 17 και το Δεκέμβριο του 2018. Δεν μπορώ να περιγράψω την χαόδη διαφορά μεταξύ της διεξαγωγής αυτών των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Και θα πάω μέσα στην ερώτηση που είναι ουσιαστικότατη αυτή τη στιγμή. Τώρα που έχετε επαρκή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο σας Προφανώς θα μπορούσατε να προχωρήσετε γρήγορα προς την ε, εκλογική μεταρρύθμιση που είχε προταθεί και ήταν επιτάπητος και η οποία όμως απέτυχε αμέσως πριν τις εκλογές ε, με δραματικές επιπτώσεις για το πρώην κυβερνών κόμμα. Ε, θα αποσύρετε κάποιες εκλογικές περιφέρειες από το σύστημα για να προχωρήσετε σε ένα αναλογικότερο σύστημα. Επίσης το 30% της ποσόστοσης του φύλου θα το εισαγάγετε και επίσης έχετε αξιόπιστη αντιπολίτευση με τόσο ισχυρή πλειοψηφία που έχετε μετά την νίκη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Χάιντε, και ευχαριστούμε για την πολύ καλή δουλειά της παρατήρησης των εκλογών. Τσάλτ Τάνεγκ για την τελευταία λέξη. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως να μην είναι 29 Μαρτίου, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει. Ε, τώρα να καλασορίσω και εγώ τον Πρωθυπουργό και να συγχαρώ για την ε, πραγματικά δημοκρατική διαδικασία της οποίας ε, ε πρωταγωνίστησε και εγώ υπήρξα αντιπρόεδρος στην προηγούμενη θητεία των, της ομάδας φίλων της Αρμενίας και πάντοτε χρειαζόμασταν μία σχέση σε πλαίσιο ΣΥΠΑ ενισχυμένης συμφωνίας διαβάζω στον τύπο ότι περιμένετε ίσως ε, κάποιες καλύτερες σχέσεις με τον Μπακού, με το Αζερμπαϊτζάν ε, και επομένως το επόμενο ερώτημά μου, κάτι που πάντα με ενδιέφερε πολύ ζωηρά, τι γίνεται με τα κλειστά σύνορα με την Τουρκία, υπάρχει κάποια περίπτωση να επιληθεί αυτό το θέμα. Αυτή την εξαιρετικά άδικη βέβαια κατάσταση όπου συνεχίζει να κλείνει τα σύνορά της η Τουρκία επί τη βάση της σχέσης της με το Αζερμπαϊτζάν και μένοντας ε, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ε, συχνά ε, πρόσφατα έφαγα με τον πρόεδρο της Γεωργίας, χώρα με την οποία πάντοτε είχαμε κάπως δύσκολες σχέσεις ως προς τις, τα δικαιώματα της αρμενικής μειονότητας. Δεν ξέρω αν έχουμε και προς αυτή την κατεύθυνση κάποια πρόοδο. Και τέλος, πάντοτε επίσης με ενδιαφέρει ιδιαίτερα εν ώψη της εκπεφρασμένης θέσεις του Τραμπ να αποσυρθεί από την JCPOA, τη σχέση με το Ιράν, η χώρα με την οποία έχετε ε, μια χερσαία οδό, επικοινωνία, σύνορα δηλαδή, ε, και με βάση τις παραδοσιακές σας σχέσεις με τη μεγάλη αρμενική κοινότητα που έχετε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς τοποθετήσετε ως προς τις κυρώσεις ε, του Ιράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Πρωθυπουργέ, πάνω από 12 συνάδελφοι πήραν το λόγο. Και τώρα εσείς ε, καλείστε να απαντήσετε όσες ερωτήσεις επιθυμείτε. Και σε 15 λεπτά θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι βουλευτές. της Επιτροπής Εκτορικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ στις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να κάνω μία ομοδοποίηση σε τρεις κατηγορίες ε, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Σε ό,τι αφορά καταρχάς τις εσωτερικές διεργασίες στην Αρμενία. Όπως είπα και προηγουμένως, είμαι βέβαιος ότι η δημοκρατία είναι καθοδόν στην, στην Αρμενία, αλλά θα πρέπει να την ενισχύσουμε, να την ενισχύσουμε με, θεσμικά, με τα θεσμικά όργανα. Και θα πρέπει φυσικά να συνεχιστούν μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό σύστημα. Αυτό θα το κάνουμε. Και προς την κατεύθυνση αυτή είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Χαίρομαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει την Αρμενία στην ε, διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Να τονίσω με πάσα ειλικρίνεια ότι προτιθέμεθα να εφαρμόσουμε πλήρως τη ΣΕΠΑ γιατί θεωρώ ότι συνάδει απόλυτα με την τρέχουσα ιστορική μας ατζέντα και με τις φιλοδοξίες μας άλλωστε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δραστηριότητες καταπολέμησης της διαφθοράς, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις για μας. γιατί θα πρέπει να καταστεί πραγματικότητα το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Είναι αδύνατον να συμβεί αυτό χωρίς την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και ναι, έχουμε διάσημες ε, υποθέσεις ε, για εγκλήματα πρώην αξιωματούχων της κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Τα δικαστήρια πλέον θα αποφανθούν για το τι μελιγενέστε. Οι δικαστές μα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποια θα είναι η μοίρα των υποθέσεων αυτών. Είναι σημαντικό, όπως ξέρετε, να υπογραμμίσουμε ότι είναι κρίσιμη σημασία η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Ξέρετε ότι ευθύ εξ αρχή εγώ προσωπικά αρνήθηκα να συνεχίσω την πρακτική που κλειδοδότησα για να λαμβάνονται δηλαδή οι δικαστικές αποφάσεις στους κόλπους της κυβέρνησης και ουσιαστικά να μεταφέρονται προς το δικαστικό σώμα. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι απόλυτα αποπισμένο για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος στην Αρμενία. Δεν είμαι βέβαιος ότι οι προηγούμενες ολιγαρχίες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ε, είχαν μοχλούς στη διάθεσή τους για να ασκούν πίεση στο δικαστικό σώμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς προτιθέμεθα να παρέμβουμε στα εσωτερικά των δικαστηρίων. Αυτό που σημαίνει ωστόσο είναι ότι θα κάνουμε πραγματικέ μεταρρυθμίσει προκειμένου το δικαστικό μα σύστημα να είναι πραγματικά ανεξάρτητο και ελεύθερο. Ακούσαμε μία ερώτηση για την ανάκτηση κλαπέντων αδικημένων. Πολύ σημαντικό το, σύστημα, το, το στοιχείο αυτό και υπολογίζουμε στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς ε, αποτελεσματικής ε, συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έγινε μια πρόταση από τον Άουσα να υποστηριχθούν ε, για να υποστηριχθεί η κυβέρνηση της Αρμενίας σε ό,τι αφορά τα κλαπέντα αυτά αντικείμενα. Για τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει πραγματικά στρατιωτική λύση για τη σύγκρουση αυτή. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σωστή ευνοϊκή ατμόσφαιρα για την εξέβρεση ειρηνική λύσεω. Ε, από την αρχή η κυβέρνησή μα έχει καταπιαστεί με το θέμα αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτό το ευνοϊκό κλίμα. Το Σεπτέμβριο έγιναν ανεφρεγμένων δηλώσεις ε, στο κοινοβούλιο μας ε, ότι οποιαδήποτε επίλυση του ζητήματος του Ναγκορνό Καραμπάχ θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το λαό της Αρμενίας, από τον Ναγκορνό Καραμπάχ και από το Αζερμπαϊτζάν. Πραγματικά ήταν ανευπροηγουμένου αυτές οι δηλώσεις από πλευρά του Πρωθυπουργού της Αρμενίας για τα δεδομένα τουλάχιστον των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ελπίζω μετά την δήλωσή μου αυτή να γίνουν και αντίστοιχε δηλώσεις από πλευρά του Προέδρου του Αζερβαϊτζάν. Δυστυχώς, ωστόσο, η ελπίδα αυτή ήταν φρούδα. Αντιθέτως, λαμβάνουμε μηνύματα από πλευράς του Αζερμπαϊτζάν για τη χρήση βίας για την επίλυση του ζητήματος χωρίς να λεφτούν υπόψη τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού του Ναγκόρνο Καραμπάχ και των Αρμενίων. Εγώ αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να διανοηθούμε οποιαδήποτε επίλυση, ταχεία επίλυση του ζητήματος. Προκειμένου να υπάρξει η λύση θα πρέπει το Αζερμπαϊτζάν να επιδείξει διάθεση διεξαγωγή διαλόγου. Δυστυχώ όμω αυτό δεν παρατηρείται στην παρούσα φάση. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ο μορφότυπο τη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ξέρετε ότι η διεθνή κοινότητα αναγνωρίζει το γεγονό ότι η σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ ε, περιέχει τρει πλευρέ: τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Και αυτό αναγνωρίστηκε διεθνώς το 1984 στην Βουδαπέστη. Έως τώρα όμως, το τραπέζι διαπραγματεύσεων το κατέχουν δύο μόνο πλευρέ. Η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν κάνουν διαπραγματεύσει χωρί τον Αγκορνό Καραμπάχ. Το πρόβλημα όμω είναι ότι οι προηγούμενοι ηγέτε τη Αρμενία ήταν από τον Αγκόρνο Καραμπάχ και ενδεχομένω να είχαν την εντύπωση ότι μπορούν να εκπροσωπούν και τον Αγκόρνο Καραμπάχ για το λόγο αυτό. Εγώ όμω δεν έχω καταγωγή από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Είμαι πρωθυπουργό της Αρμενία. Δεν είμαι πρωθυπουργό του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο λαό ε, του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν συμμετέχει στι αρμενικέ εκλογέ. Δεν είναι πολίτε της Αρμενία. άρα δεν είμαι σε θέση να διαπραγματευτώ εξ ονόματος του Ναγκορνό Καραμπάχ, μόνο εξ ονόματο τη Δημοκρατία τη Αρμενίας. Άρα το δεύτερο βήμα είναι να δημιουργηθεί ένα σωστός μορφότυπος για την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων προκειμένου προκειμένου να γίνουν ουσιαστικέ διαπραγματεύσεις. Και θα ήθελα να επιμείνω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν χωρίς την συμμετοχή του Ναγκόρνου Καραμπάχ στην όλη αυτή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία τώρα. Ξέρετε, το θετικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέτει γεωπολιτικούς όρους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Αρμενία. η ατζέντα συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πλήρης μεταρρυθμιστική ατζέντα που περιλαμβάνονται στην ΣΕΠΑ και θα υλοποιηθεί 100%. Ασφαλώς, οι σχέσεις μας με τη Ρωσία είναι πολύ σημαντικές για μας και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Το μεγαλύτερο τμήμα της ε, συνεργασίας μας έχει να κάνει με την Οικονομική Ένωση και την ε, ατζέντα για την ασφάλεια. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε διαφανείς για αμφότερες τις σχέσεις αυτές. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία συνωμοσία κατά της Ρωσίας στις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε αντίστοιχα υπάρχει οποιαδήποτε συνωμοσία για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Φυσικά η συνεργασία θα πρέπει να διέπεται από ένα βαθμό ενέργειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το θέμα της ενέργειας προφανώς είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας έχουμε συνεργασία και με το Ιράν και σκοπεύουμε να εξελίξουμε τις σχέσεις μας και με το Ιράν. Προσφάτως επισκέφτηκα το Ιράν. Συζητήσαμε τις δυνατότητες μεταξέλιξης της σχέσης μας σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Ό,τι αφορά τώρα τα συγκεκριμένα βήματα. Γνωρίζετε ότι η δική μας η ιδεολογία είναι η ίδια. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και τις οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις. Ποια ήταν άλλωστε η βασική ιδεολογία για τις οικονομικές μας μεταρρυθμίσεις. Να ενθαρρύνουμε τον κόσμο στη τελική ανάλυση, να κάνει συγκεκριμένα βήματα και να πάρει το μέλλον του στα χέρια του. Από πλευράς οικονομικών αλλαγών και οικονομικής ε, επανάστευσης θα ενθαρρύνουμε το λαό μας να αποδεθεί σε οικονομικές δραστηριότητες. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί πριν από την ε, Επανάσταση είχαμε ολιγαρχίες, μονοπόλια. Όλα αυτά περιόριζαν τις ευκαιρίες οικονομικής δραστηριότητας. Πλέον λοιπόν έχει ανοίξει το πεδίο δράσης και τώρα θέλουμε να υπάρχουν ίσοι όροι για όλους. Θα μεταρρυθμίσουμε τον φορολογικό μας κώδικα. θέλουμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πεδίο στην οικονομία μας, την μικροοικονομία για να απελευθερώσουμε τον κόσμο αυτόν από το βάρος το, της φορολόγησης και θέλουμε να κάνουμε και ρυθμιστικές ελαφρύνσεις για να καταστούν πιο εύκολες οι επενδύσεις, να καταστούμε πιο ευνοϊκοί και ελκυστικοί για επενδύσεις. για την ανάπτυξη των υποδομών και το καθεξής. Mm. Και δυστυχώς βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος ομιλίας μου για την ατζέντα αυτή στο σύνολό τη. Προφανώς και χρειάζεται τεχνική και οικονομική αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ενδεχομένως και συμβουλαστική ε, για να καταστεί πιο δυνατή, πιο στεναρή η δημοκρατία μας από οικονομικής, πολιτικής και τεχνικής άποψης, αλλά για μένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Αρμενία έχουν εγκαθιδρυθεί μόνιμα. Δεν θα υπάρξει πίσω γύρισμα σε διεφθαρμένα καθεστώτα. Ευχαριστώ πολύ. Prime Minister Pashinyan. Πρωθυπουργέ Πασινιάν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων των συναδέλφων ε, που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Πάρα πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω να έχετε εδώ καλή συνέχεια και γόνιμη συνομιλία στις Ευχαριστώ πολύ. We would like to continue our meeting. If the Armenian... Λοιπόν, παρακαλώ την αρμενική αντιπροσωπεία να έχει την καλοσύνη να βγει από την αίθουσα. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολύ χώρο απ' έξω να δώσετε όλες τις συνεντεύξεις που θέλετε. So, ladies and gentlemen, I would like... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Καθίστε όμως παρακαλώ για να αρχίσουμε. You either leave room or you're seated. Λοιπόν, είτε θα καθίσετε είτε θα βγείτε. Ένα από τα δύο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. we obviously still have a number of friends of Armenia leaving Βλέπουμε της Αρμενίας να αποχωρούν ακόμα μερικοί. So, we continue our meeting with... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το σημείο υπαριθμών 7. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, υπάτη πρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με το πεδίο εφαρμογή και την εντολή για τους ειδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτρια είναι η κυρία Βάουτμανς, η οποία απουσιάζει. EPP group Παρακαλώ τα πηγαδάκια του ΕΛΚ να σταματήσουν. Έτσι κι έχει πέρασει η ώρα και θα ψηφίσουμε. Αποουσιάζει η συγγήτρια, οπότε θα περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Έχει κανείς να πει τίποτα, όχι. Ωραία. Προχωρούμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 22. Α, συγγνώμη, κυρία Νίνα Γκίλ, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περίμενα να είναι εδώ η συγκήτρια. Απουσία της συγκήτριας λοιπόν. Θέλω να πω στους κοιόδες ότι έχω μια ε, προφορική τροπολογία που έχει κυκλοφορήσει. Όταν φτάσουμε στο σημείο N, ε, ε, παρακαλώ μου δώστε το λόγο για να σας παρουσιάσω την προφορική μου τροπολογία. Οπωσδήποτε και σας ευχαριστώ. Σας βλέπω αναστατωμένους. Δεν ξέρω τι γίνεται, συνάδελφοι. Ε, καθίστε για να ψηφίσουμε. Λοιπόν, η τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές, αυτό θέλει έλεγχο σας παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε. Την τροπολογία 36 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα ή δεν θέλουν να ψηφίσουν, πας περιπτώσει πέρας. Εγκρίνεται 29-21. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 καταπίπτει, 41 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ φωνές από κάτω. Τη 42 θέλετε να ελέγξουμε μάλιστα αρχίζει τώρα. Ε, excuse me, Δύο ΕΛΚ υπεράριθμοι. Καλά, ποτέ έτσι κι αλλιώς δεν είναι αρκετοί οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ, αλλά αυτή τη στιγμή περισσεύουν δύο. Μπορείτε να το λύσετε αυτό σας παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίθηκε 29-16. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, ε, 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 67 αρχής τώρα η ψηφοφορία. 67. It's okay. The vote is closed. This has been rejected. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 70 καταπίπτει, συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Παρακαλώ, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία παριθμών 72. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές. Ορίστε. Θέλετε έλεγχο για την 74. Παρακαλώ, αρχίζει τώρα. Κύριε Γιούρεκ, δική σας είναι. Πέρας. Ω, καταπορρίφθηκε. Και τώρα πάμε στην 78 και είναι η ώρα της Νίνα, στο σημείο M και όχι N. Ε, Κυρία Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορεί να γνωρίζετε ότι την περασμένη εβδομάδα ορίστηκε νέος ενδεταλμένος ο Γκίλμορ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις 28 Φεβρουαρίου είχαμε τα αποτελέσματα του Συμβουλίου που διεύρυναν την εντολή του από τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και στη Διεθνή Ποινική Δικαιοσύνη. Δεδομένου αυτών των εξελίξεων, λοιπόν, θα ήθελα να τροποποιήσω την αρχική μου τροπολογία, υπαρίθμη 78, με μια προφορική, η οποία έχει κυκλοφορήσει ε, και την έχουν στα χέρια τους οι συνάδελφοι. Αλλιώς να σας τη διαβάσω. Μπορώ, αν θέλετε. Αλλιώς να την ψηφίσουμε, Πρόεδρε, αν την έχετε. Εξαιρετική προφορική τροπολογία αυτή, ψήφι υπέρ, κατά, θαυμάσια εγκρίθηκε και προχωρούμε. 81. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές έλεγχος. ελέγχουμε το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 81. Ελεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά αποχές την ε, ελέγχουμε. 88 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 89 υπέρ, κατά αποχές Πάλι έλεγχο και για την 89 χρειαζόμαστε. Αρχίζει τώρα η επαλήθευση. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 91 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 97 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος επελθεύουμε τώρα την 97 αρχής ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές. Έλεγχος της 98 αρχίζει τώρα. Πέρασε. Απορρίπτεται. 99 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ετιολογικές σκέψεις 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται, άραγε. Ας την ελέγξουμε για καλό και για κακό. Τη 13 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Νταλούνται. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολόγια 14 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ φωνάζει ο κύριος Τάνοκ. Αρχίζει λοιπόν η ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 20. Γιατί λείπουν συνέχεια τρεις συνάδελφοι, δεν ψηφίζουν δηλαδή. E too much in the moment. Ακόμα περισσεύει ένας από το ΕΛΚ αυτή τη στιγμή. Πέρας. Απερίφθη Τσάρλς, τι να κάνουμε τώρα, 10.41. Αυτή και αν ήταν ψηφοφορία κρίσιμη. 21 είπε, κατά αποχές εγκρίθηκε. Αιτιολογικές αναφορές τώρα. 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές 4. Έλεγχος ηλεκτρονικός αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 6 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία πέρασε εγκρίθηκε 7 υπέρ κατά αποχές και αυτό θέλει έλεγχο πάμε πέρασε εγκρίθηκε το σύνολο του σχεδίου συστάσεως όσο τροποποιήθηκε, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Πέρασα. Εγκρίθηκε. 50 ψήφοι υπέρ και 3 αποχές, χωρίς κατά. Ωραία. Προχωρούμε στο σημείο. 8 δεν έχουμε. 9 πρωτόκολλο τη Ευρωμεσογειακής Συμφωνία σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών του Αφενό και του κράτου του Ισραήλ αφετέρου ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση τη Δημοκρατίας Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκητής ο Πρέντα δεν θέλει το λόγο. Μπορούμε να περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ είναι μία ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίθηκε 47 υπέρ, μία ψήφος κατά. Ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών ΑΦΕΤ και το επόμενο θέμα είναι κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού θέσπιση μηχανισμού γειτονίας ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Μην φεύγετε τα μέλη της ΑΦΕΤ όσο φτάνουν οι συνάδελφοι της Έχουμε και αύριο 5 μέχρι το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΦΕΤ και κλεισμένων των θυρών για ανταλλαγή απόψεων με την ΕΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση στην Αλβανία και η επόμενη τακτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου. Πριν κηρύσω τη λήξη της Επιτροπής ΑΦΕΤ έχουμε τίποτα στα διάφορα. Όχι. Καλωσορίζω όλα τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ και ιδιαίτερα την πρόεδρο τη Λίντα Μακάβεν. Καλώς όρισες. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε απευθεία με την ψηφοφορία, αν συμφωνείτε. Το σύστημα είναι έτοιμο. Εγώ θα προεδρεύσω ή η Λίντα.